Good afternoon, my dear colleagues. Um, I start with the... Γεια σας. Ξεκινάμε με τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις του Προέδρου. Καλώς ήρθατε μετά από τις διακοπές. Η ελπίδα μου είναι ότι έχετε ξεκουραστεί όλοι και ανανεωμένοι και έτοιμοι για τις συνεδρίες της Επιτροπής μας. Η ημέρησια διάταξή σας έχει σταλεί ήδη από τα τέλη Αυγούστου και είναι στο φάκελό σας θα, δει, θα μεταδοθεί και στο διαδίκτυο αυτή η συνεδρίαση και θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά στη διαδικασία ψηφοφορίας, οπότε μετά από την ακρόαση των τριών υποψηφίων για το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να έχετε την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας μαζί σας. Τα εξής πρακτικά έχουν δημοσιευθεί της 4 Ιουλίου 2016 και 13-14 Ιουλίου δεν έχουμε λάβει ακόμα ενστάσεις σε σχέση με τα πρακτικά. Ελήψη πρακτικών μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Και επειδή έχουμε πολύ φορτωμένη σε διάταξη, θα έλθω στο θέμα της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του ελεκτικού συνεδρίου και με μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω εδώ τον κύριο Λαζάρου Όταν σας βλέπω σκέφτομαι τα θέματα της απαλλαγής, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ανανέωση της εντολής σας και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Ιγκόρ Σόλτζος, ο οποίος είναι ο εισηγητής μας για τα θέματα αυτά. Σας δίνω το λόγο και παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε κάποια σχόλια. Καταγράφω αυτούς που θέλουν να θέσουν ότι κύριε Σόλτζος έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. έχουμε επανέλθει στον σωστό δρόμο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και εγώ βλέποντας τον κύριο Λαζάρου σκέφτομαι τις δημόσιες προμήθειες και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος του ελεκτικού συνεδρίου για τα θέματα αυτά. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν θα ήθελα να παρουσιάσω τον υποψήφιό μας. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερα καινούριο να σας πω για τον κύριο Ζάρου. Φυσικά ξέρετε ότι ήταν μέλος του ελεκτικού συνεδρίου από το 2010. Ήταν από το 2005-2015 έως 2005-2010. Επίσης υπήρξε αρμόδιος ε, υπεύθυνος για τα θέματα εσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1999 από το 2005. 2015 εως 2005 2010 επισης υπηρξε αρμοδιος υπέρ για τα θεματα εσοδων εργαστεί στον ε, ιδιωτικό τομέα περαιτέρω. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις δείτε στο βιογραφικό του. Κατόπιν όλων αυτών λοιπόν και έχοντας ελέγξει το βιογραφικό του και γνωρίζοντας πολύ καλά το έργο του ως ε, μέλους του Ελεκτικού Συνεδρίου μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε καμία ανησυχία σε σχέση με την ανεξαρτησία του ή την ικανότητα και τα καθήκοντα τα οποία έχει αναλάβει στο παρελθόν. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά τα τελευταία χρόνια με το τμήμα του στο ελεκτικό συνέδριο. Πιστεύω λοιπόν ότι ίσως είναι καλύτερα να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Λαζάρου για να παρουσιάσει την δική του θέση και τις απόψεις του για το μέλλον. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Σεϊτέ, να σα συνεχίσω στα ελληνικά, στην μητρική μου γλώσσα και θα απαντήσω μετά στι ερωτήσει στα αγγλικά. Πρόεδρε, κύριε εισηγητή, έντιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχοντας προταθεί από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι τιμή μου που παρουσιάζομαι ενώπιον σας για να ζητήσω τη θετική σας γνώμη και αυτή της Ολομέλειας για να διοριστώ μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για δεύτερη θητεία. Από το διορισμό μου τον Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο 2014 υπηρέτησα στο τμήμα 1 και ακολούθω στο τμήμα 2 τα δύο αυτά τμήματα είναι αρμόδια για τις δαπάνες της επιμερισμένης διαχείρισης. Ήμουν εισηγητή για αριθμό ειδικών εκθέσεων επίτευξη αποτελεσμάτων και ο εκπρόσωπο και των δύο τμήματων στο οριζόντιο τμήμα ΚΑΤ. Από το Φεβρουάριο 2014, μετά από αίτημα του Προέδρου του Συνεδρίου και των συναδέλφων μου, ανέλαβα ως το αρμόδιο μέλος για τη δήλωση αξιοπιστίας επί των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον ω μόνιμο μέλος του τμήματος ΚΑΤ. Είμαι υπεύθυνο για το συντονισμό των εργασιών που σχετίζονται με την ετήσια έκθεση μα και για τη διασφάλιση τη συνοχή και τήρηση τη μεθοδολογία ελέγχου του συνεδρίου στην υποκείμενη εργασία για την δήλωση αξιοπιστίας. Είμαι εισηγητής, μεταξύ άλλων, για τα κεφάλαια της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τη δήλωση αξιοπιστίας και τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση. Η υπηρεσία μου στο συνέδριο μου επιφέρει ευπρόσδεκτες προκλήσεις και επαγγελματική ικανοποίηση. Τέτοιες προκλήσεις περιλαμβάνουν πρώτον περαιτέρω βελτίωση της επικοδομητικής επαγγελματικής μας συνεργασίας με την Επιτροπή σας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω συστηματικής ανταλλαγής απόψεων. Δεύτερον, δέουσα προσοχή στα ενδιαφέροντα και ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών στον προγραμματισμό του ελέγχου μας περιλαμβανουμένου πρωτοβουλειών για συγκεκριμένη πληροφόρηση ανακράτος μέλος ή γεωγραφική επισκόπηση. Τρίτον, σταδιακή εξέλιξη της ετήσιας μας έκθεσης ως ένα εργαλείο με περισσότερη προστιθέμενη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τέταρτον, εξέβρεση κοινή αντίληψη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιμέτρηση λαθών στις δημόσιες συμβάσεις. Φυσικά, παρόλο που ο ελεκτής και ο ελεγχόμενος δεν θα συμφωνήσουν σε όλα τα θέματα, η κοινή αντίληψη είναι πάντα υποφελής. Και πέμπτον, καθορισμό ενωρίτερη ημερομηνία δημοσίευση τη ετήσια μα έκθεση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνεισφορά στη διασφάλιση επίτευξη αυτού του στόχου. Σε συνεννόηση με την Επιτροπή σα, η ετήσια έκθεση 2015 θα δημοσιευθεί και παρουσιαστεί σε εσά στις 13 Οκτωβρίου, περίπου ένα μήνα νωρίτερα από προηγούμενα. Και επαγγελματική ικανοποίηση γιατί, πρώτον, μου αρέσει η δουλειά μου, τόσο η τεχνική πλευρά όσο και η επαφή με συναδέλφους, την Επιτροπή σας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, Ειδικότερα προσβλέπω στη συνέχιση της ανταλλαγής απόψεων μαζί σας για τα επόμενα βήματα στην εξέλιξη της ετήσιας έκθεσης. Δεύτερο, είχα την ευκαιρία να αποκτήσω πολύτιμη εμπειρία σε όλο το φάσμα των εργασιών του συνεδρίου. Τρίτο, συμβάλλω στην παραγωγή εκθέσεων σχεδιασμένες να υποβοηθήσουν τις αρχές προϋπολογισμού και χορήγησης απαλλαγής στην άσκηση των καθηκόντων τους για έλεγχο. Επιπρόσθετα από τις αξίες που ανέφερα νωρίτερα, ήμουν εισηγητής και από τη γνώμη του συνεδρίου επί της πρότασης κανονισμού για το ΕΦΣΥ και τέταρτο γιατί αισθάνομαι ότι η συμβολή μου στις εργασίες του συνεδρίου εκτιμάται και αναγνωρίζεται ευρέως. Με την αναδιοργάνωση του συνεδρίου σε οργανισμό με προτεραιότητα δράσεων στις αρχές Ιουνίου το τμήμα ΚΑΤ έγινε τμήμα 5 αναλαμβάνοντας μέρος της δουλειά του ΚΑΤ και του τμήματος 4. Η κύρια θεματική αρμοδιότητα του τμήματος 5 στο οποίο εκλέγηκα πρόεδρος και με αυτή την ιδιότητα μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, είναι η χρηματοδότηση και διοίκηση της Ένωσης. Το τμήμα 5 είναι επίσης το συντονιστικό τμήμα για την ετήσια έκθεση και μετά από απόφαση του συνεδρίου συνεχίζω με τα ίδια καθήκοντα ως μέλος για την ετήσια έκθεση εισηγητής για το κεφάλαιο της δήλωσης αξιοπιστίας. Επιπρόσθετα, είμαι εισηγητής για την ειδική έκθεση που προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τον Νοέμβριο σχετικά με τη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη γνώμη του συνεδρίου επί της επικείμενης πρότασης της Επιτροπής για αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προϊόντα και τα επιτέγματα μας είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Είμαι ευτυχής που έχω τη συνεισφορά και τη συμπαράσταση των συναδέλφων μελών του συνεδρίου της ομάδας μου και του προσωπικού μας, όπως επίσης και τη συμπαράσταση και κατανόηση της συζύγου μου και της οικογένειάς μας. Τους ευχαριστώ όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο σημαντικές προκλήσεις. Αυτό απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτευχθούν πιο χειροπιαστά αποτελέσματα στη διαχείριση του προϋπολογισμού. Αυτά περιλαμβάνουν επίτευξη των πολιτικών στόχων που να έχουν εμφανή αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών, κάνοντας κάθε ευρώ που δαπανάται να μετράει με ταυτόχρονη τήρηση των κανόνων και κανονισμών των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και με προσήλωση στις κοινωνικές αξίες και την ηθική. Ως ελεκτής θα συνεχίσω να είμαι ανεξάρτητος, σταθερός αλλά δίκαιος και επικοδομητικός, με κριτική όταν χρειάζεται, αλλά με ενθάρρυνση και υποστήριξη όταν απαιτείται. Προσβλέπω τώρα στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς. Τα καταφέραμε αλλά τα προβλήματα. Ευχαριστώ και την τσέχη Διερμηνία. Λοιπόν, ένας ε, προς τις ερωτήσεις. Η κυρία Αγιάλα Σαντέρ, ε, έχει πρώτη τον λόγο για ερωτήσεις. όχι και εγώ τις δικές μου, αλλά δίνω πρώτα τον λόγο στα μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τη γραμματεία, όλα, όλους αυτούς που είναι παρόντες. Καταρχήν να τους ευχηθώ καλό φθινόπωρο μετά από ένα ευχάριστο καλοκαίρι και ελπίζω ότι έχουν ανακτήσει τις δυνάμεις τους γιατί η οικοδόμηση Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτήσει όλες τις δυνάμεις μας. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχουμε ενωπιών μας είναι αυτή η ανανέωση των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου και ο κύριος Λασάρου, τον οποίο χαιρετίζω, το γνωρίζω πολύ καλά. Έχουμε εργαστεί πολύ ευδοκίμως μαζί σας για θέματα και εύκολα και δύσκολα, ιδίως σε σχέση με την ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και τις διάφορες εναλλακτικέ οδούς για το μέλλον του ελεκτικού συνεδρίου. Πάντα είχατε ένα επικοδομητικό πνεύμα, κρατώντας πάντα μια στεναρή στάση από τη δική σας πλευρά, αλλά με τη δυνατότητα να ακούτε πάντα τις απόψεις των άλλων να μπορείτε να εξετάζετε και να διερευνείτε και άλλες δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Είπατε σαφώς ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει λάβει υπόψη τις δικές μας θέσεις ότι θα πρέπει να προσεγγίσει περισσότερο στις προγραμματικές του δηλώσεις στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο σε αυτά τα οποία προσπαθούν να επιτύχουν τα μεγάλα θεσμικά όργανα του Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Θα σας ρωτήσω αν έχετε κάποια ιδέα για το πώς μπορείτε να προσεγγίσετε περισσότερο αυτό το θεματολόγιο χωρίς φυσικά να υπονομεύσετε την ε, ανεξαρτησία του ελεκτικού συνεδρίου αλλά να δράτε λιγάκι εξάντε για να προωθήσετε αυτά τα θέματα. Ένα δεύτερο θέμα που έχει να κάνει πάλι με την προσέγγιση του ελεκτικού συνεδρίου από την ε, αξιο... προς την αξιολόγηση επί τη βάση των αποτελεσμάτων <clears throat> για την εφαρμογή του προπολογισμού. Θα ήθελα να σας ε, θέσω το εξής ερώτημα αν πιστεύετε ότι το ελεκτικό συνέδριο, όπως είναι σήμερα οργανωμένο, έχει αρκετούς πόρους, αρκετές ικανότητες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις εκθέσεις αυτές επί των αποτελεσμάτων που να είναι πραγματικά αμερόληπτες. Να μην δίνουν την εντύπωση ότι έχουν πολιτικό χαρακτήρα, ότι εκφράζουν ανάχα την πολιτική άποψη κάποιου μέλους του ελεκτικού συνεδρίου, όπως κάποιες φορές στο παρελθόν είχαμε την εντύπωση, αλλά είναι εκθέσεις οι οποίες εξετάζουν πραγματικά τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, κάτι το οποίο δεν είναι βέβαια λογιστικό και μόνο σε σχέση με την εφαρμογή του προπολογισμού. Και συγχρόνως αυτές οι εκθέσεις θα πρέπει να έχουν αυτήν την απόλυτη ουδετερότητα και την αμεροληψία σε σχέση με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Τρίτο, και πάλι για την ετήσια έκθεση. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Από τη μία πλευρά είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψουμε αυτό το οποίο έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα και ήταν ένας από τους πυλώνες της διαδικασίας αυτής, η ετήσια δηλαδή η απαλλαγή που χορηγείται από το Κοινοβούλιο Έχουμε κάποια θέματα τα οποία δημιουργούν πολλές ε, απαιτήσει για μας, όπως είναι η κρίση των προσφύγων, τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, συν τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειάζεται κάπως να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η πληροφορία στην ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Γιατί η κοινή γνώμη, οι πολίτες της Ευρώπης δεν μπορούν να έχουν την εντύπωση ότι όλα πάνε στραβά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο προπολογισμό δεν λειτουργεί και γίνονται μοναχα και ατασταλίε, όταν η πραγματικότητα είναι ότι λειτουργούν, υλοποιούνται τα διαφορετικά ταμεία και τα διαφορετικά προγράμματα, μερικέ φορέ με καθυστέρηση βέβαια, αλλά πιστεύω ότι εξακολουθούμε να είμαστε μια περιοχή όπου υπάρχει πραγματική ανάπτυξη, υπάρχει σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχει η κατάλληλη μέρημνα για τα κοινωνικά θέματα στο μεγαλύτερο μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει αυτό πρέπει να το κατανοήσουν και οι πολίτε μας. Δεν ξέρω λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό, γιατί αυτό είναι από τα θέματα όπου εσεί έχετε σταθεί πρωτοπόρο, πιστεύω. Ο κ. Λαζάρου. Κύριε Γελασέντερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όντως, το ελεγκτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο, εξωτερικός ελεγκτής των θεσμικών οργάνων. Μέσω των εκθέσεών μας προσπαθούμε εργαζόμενοι σκληρά να βελτιώσουμε την λογοδοσία εν γέννη ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ναι, σημειώσαμε στην τελευταία μας ετήσια έκθεση ότι δεν εστιάζουμε επαρκώς σε θέματα απόδοσης. στην απόδοση των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή και στο γεγονός επίσης ότι τα προγράμματα που συνομολογούν τα κράτη-μέλη με την Κομισιόν δεν συνάδουν ε, επαρκώς με τους στόχους του 2020. Έχουμε τονίσει ότι υπάρχει έλλειψη εστίαση σε θέματα απόδοσης. Και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναφώς να αλλάξει τη συνήθεια στην νοοτροπία και εντός της Κομισιόν και στα κρατημέλη μελη για να τονιστεί ακόμη περισσότερο η ανάγκη να, να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Το ελληνικό λοιπόν συνέδριο και εγώ προσωπικός ανέκαθεν προσπαθούσαμε να έχουμε τακτικές επαφές και ανταλλαγές απόψεων με τους εμπλεκομένους και δει με την Επιτροπή σας, την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες σας κατά τη διενέργεια των ελέγχων μας. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πεπερασμένους πόρους στη διάθεσή μας, πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες, να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες μας και έτσι λειτουργούμε με στόχο όχι μόνο την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης αλλά και των ειδικών εκθέσεων που έχουν και ίσως περισσότερη αξία στους συγκεκριμένου εμπλεκομένους και δει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας. Έτσι, χειριζόμαστε θέματα που, έχουν, που άπτονται του προπολογισμού αλλά και που ενδιαφέρουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Αναφερθήκατε στο κατά πόσον πρέπει να επανεφεύρουμε τον τρόπο, να επανασχεδιάσουμε τον τρόπο δημοσίευση των ετησίων εκθέσεων. Ξέρετε, ε, αυτό γίνεται λαμβάνοντας υπόψη, όπως ε, προείπα, τα συμφέροντα και τι ανησυχίε όλων των εμπλεκομένων και βεβαίω των Ευρωπαίων πολιτών. Τι προσπαθούμε να κάνουμε με τι εκθέσει μα και με την ετήσια έκθεσή μα, ακόμη περισσότερο. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε το δικαίωμα έγκαιρης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων αυτών που ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα, ελέγχου, που εμπλέκονται στα θέματα προπολισμού, για να βελτιωθεί εν γέννη η διαχείριση των δημοσιονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαρδαμά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαζάρου, ευχαριστώ με τις ευκαιρίες για να δηλώσω ότι η συνεργασία μας ήταν εξαιρετικά ευχάριστη και ομαλή. Ήσασταν ε, ιδιαίτερα ανοιχτό και ειλικρινής επί όλων των θεμάτων στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την Επιτροπή μας. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, λεγόμενες ε, αναχώρα συστάσεις. Ε, πώς μπορούν να βελτιωθούν, να αναπτυχθούν περαιτέρω κατά τη γνώμη σας. Και δεύτερον, δεδομένου ότι είστε υπεύθυνο πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης πριν από λίγα χρόνια όσον αφορά την γεωργία και την συνοχή από το 2007 στο 2013 τα σχετικά ε, στοιχεία είχαμε μια εξαιρετική έκθεση που διαβάσαμε το 2014 στοιχεία αναχώρα με πολύ άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία γενικά για το θέμα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση λοιπόν ως προς αυτό αυτή η πρωτοβουλία, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που αναλάβατε πώς μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω πώς μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω Ευχαριστώ κύριος Λαζάρου Ευχαριστώ κύριε Σαρβάμα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η αναχώρα πληροφορίε τα αναχώρα στοιχεία. Είναι ένα θέμα το οποίο ξέρω ότι σας ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό εσάς, την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο. Ε, προσωπικά θα αποκαλούσα τα στοιχεία γεωγραφικής φύσης ε, στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δημοσιονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να πούμε ποια χώρα τα κάνει καλύτερα ή χειρότερα. Μέσω λοιπόν αυτών των ε, γεωγραφικά προσανατολισμένων ε, στοιχείων μπορούμε να αναδείξουμε τα καλά παραδείγματα αν θέλετε, να τονίσουμε τα ισχυρά στοιχεία και να δούμε πού χρειάζεται βελτίωση. Είναι το θέμα στο οποίο Αναφέρθηκε νομίζω η κυρία Γιάννα Σέντερ λίγο πριν στην παρέμβασή τη. Έχουμε κάνει βήματα προσπαθώντας να καταλάβουμε καλύτερα τα γεωγραφικά αυτά στοιχεία για την περίοδο 7-13. Μια άλλη πρωτοβουλία είναι τα παρατήματα. Το παρατήμα είναι της έκθεσης ε, συγκεκριμένα φορά την συχνότητα των διαπιστούμενων σφαλμάτων σε κάθε χώρα όμως πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η εντολή μας δεν μας επιτρέπει να δώσουμε το ποσοστό σφάλματος αναχώρα. Αυτό το γνωρίζει η Επιτροπή σας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Όμως, ναι, συμφωνώ, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τα ε, στοιχεία αυτά αναχώρα ή αναγεωγραφική, αν θέλετε, περιοχή. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο της Κομισιόν ως επιβλέποντος και ως ελεγκτή και να ασκήσουμε περαιτέρω πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέγει πιο αξιόπιστα στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Έτσι ώστε και εμείς με τη σειρά μας να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα το έργο της Κομισιόν μέσω της ε, ετήσιες εκθέσει πεπραγμένων, η Κομισιόν κάθε χρόνο μας δίνει πολύτιμα στοιχεία αναχώρα, γεωγραφική περιοχή. Στη φάση αυτή όμω τα στοιχεία αυτά δεν είναι επαρκώ αξιόπιστα. Πρέπει λοιπόν να οθήσουμε την Κομισιόν να συλλέγει πιο αξιόπιστα στοιχεία. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα το κάνουμε, να ξέρετε, στο ελεγκτικό συνέδριο, είναι στο πρόγραμμά μας. Θα το συζητήσουμε μάλιστα τέλη Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του τυσίου στρατηγικού σεμιναρίου, όπως το αποκαλούμε. Εγώ προσωπικώς υποστηρίζω αυτά τα, τη συλλογή αυτών των στοιχείων, ανά γεωγραφική περιοχή ή χώρα. Εκεί έχω καταλήξει. Και όπως είπα θα το συζητήσουμε στο πλαίσιο της στρατηγικής μας ανταλήξης υπόψεων και θα το λάβουμε υπόψη μας στον προγραμματισμό των ελέγχων μας. Έχω και τον κύριο Σόλτες τώρα, ο οποίος θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Κύριε Λαζάρου, όλο και περισσότεροι ε, υποψήφοι για το ελεκτικό συνέδριο συμπεριλαμβάνουν τα θέματα ισότητας των φύλων και το θέμα της δεοντολογίας και της ηθικής μέσα στα πλαίσια της ε, παροχής εκθέσεων. Πού βλέπετε λοιπόν την ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να δοθεί από το δικό σας ε, θεσμικό όργανο για θέματα όπως είναι τα θέματα της ισότητος, της οικολογίας, της και ε, δεοντολογίας κτλ. Ευχαριστώ κύριε Σόλτες. βάση της συνθήκης, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε, να κάνουμε λογιστικό έλεγχο των στοιχείων που ε, αντιμετωπίζεται με τρεις επικεφαλίδες της ε, συνθήκες, οικονομία, ε, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Εμείς λοιπόν έχουμε και ένα κώδικα δεοντολογίας στον οποίο ακολουθούμε και ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα για την ε, λογιστική καταγραφή. Συγχρόνως όμως. Εξετάζουμε όμως παράλληλα το κατά πόσο υπήρξε σεβασμός των τριών ε που είπαμε προηγουμένως στα αγγλικά οικολογία, ε, ισότητα και ηθική. Έχουμε ε, δημοσιεύσει μια σειρά από ειδικέ εκθέσεις για τα θέματα αυτά. Έχουμε αναφέρει ήδη στις απαντήσεις μας στα σχόλια του Κοινοβουλίου σε σχέση με τη διαδικασία απαλλαγή. Έχουμε τονίσει ότι μια τέτοια έκθεση είναι τα θέματα των ε, τροφικών ουσιών στην Βαλτική. Αυτό καλύπτει την οικολογία. Έχουμε αντιμετωπίσει θέματα όπως είναι η ποιότητα των υδάτων, η διαχείριση των λιμάτων, αλλά οικολογικά θέματα. Έχουμε αντιμετωπίσει θέματα ισότητας, παραγωγής για την ε, για τα κονδύλια και την υλοποίηση των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου. Εγώ από τα πρώτα θέματα που αντιμετώπισα στο ελεκτικό συνέδριο ήταν η ισότητα στην κατανομή των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου. Είχαμε στο παρελθόν το θέμα της ε, δαπάνης, των δαπανών για την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών. Είχαμε επίσης μια έκθεση για την απάτη ΦΠΑ. Επομένως αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα θέματα μέσα στη φυσιολογική, στην καθημερινή μας εργασία και εστιάζουμε περισσότερο στις ειδικές μας εκθέσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λασάρ. Ο κύριος Μπαλτσίτης είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Λαζάρου είναι από τα πιο ενεργά μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου και τα έξι χρόνια που έχετε εργαστεί στο Ελεκτικό Συνεδρίο έχετε δημοσιεύσει, έχετε συντάξει εκθέσεις για τις μεταφορές, για την ενέργεια. Όπως είπατε, είσαστε ένας από τους συντάκτες της έκθεσης αυτής για τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να επέλθουν στο ελεκτικό συνέδριο. Και είστε κατά κάποιο τρόπο ο πρίτανης του πέμπτου τμήματος που ασχολείται με τα θέματα χρηματοδότησης και διοίκησης στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχετε απαντήσει όμως πλήρως το ερώτημά μου για το θέμα αυτό. Σίγουρα θα ανανεωθείτε στην, ε, στα καθήκοντά σας αυτά στο ελεκτικό συνέδριο και η ελπίδα μου είναι ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και έτσι θα μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε περαιτέρω την ανάγκη να παράγει πιο αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία η Κομισιόν, γιατί αυτό είναι και, το, και η βάση του έργου μας και στο Κοινοβούλιο και στο Ελεκτικό Συνέδριο. Πού νομίζετε ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο όμως την προσοχή μας στο μέλλον. Ποιοι είναι οι τομείς όπου θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες για την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων. Σας ευχαριστώ κύριε Παλσίτη για τις ερωτήσεις που μας κάνετε. Και όντω, πρωταρχικός στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή θα διαβιβάζει πιο αξιόπιστα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη. Φυσικά, Μπορεί η Επιτροπή να είναι τελική υπεύθυνη για την εκτέλεση του προπολογισμού, αλλά και τα κράτη-μέλη φέρουν αντίστοιχο μερίδιο τη ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν να τα ενθαρρύνουμε, να ασκήσουμε πίεση, προκειμένου να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και προκειμένου να είναι πιο αξιόπιστη η δουλειά του. Πού θα πρέπει τώρα να εστιαστούμε στο μέλλον. προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικές οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τώρα, όπως εντοπίσαμε και όπως καταλήξαμε στην έκθεσή μας του 2014, θα πρέπει να είναι η απορρόφηση των εκκορυμμένων δαπανών στα κράτη-μέλη. Το use it or lose it. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία που επικρατεί θα πρέπει να αλλάξει και εστιαστήκαμε ιδιαίτερως στο ποσοστό σφαλμάτων τα τελευταία χρόνια. Αλλά ενδεχομένως να μην εντοπίζεται και το πραγματικότερο πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα γίνονται οι πάντα με νόμιμο και σωστό τρόπο, χωρίς όμως να μην υπάρχει αδικτύπωση ό,τι αφορά τη ζωή των πολιτών. Και αυτό το τονίσαμε σε, διάφορα, ε, σε διάφορες εκθέσεις. Μία ειδική έκθεση έρευνας που αποτελεί καλό παράδειγμα της έλλειψης της νοοτροπίας αυτής που επικρατεί για ε, την απόδοση, την αποδοτικότητα. Αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, ε, το κοιτάξαμε σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για τις υποτομές των δρομείων. Θα πρέπει λοιπόν να ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει ένα πακέτο το οποίο προσανατολίζεται στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και στην ε, επερχόμενη αναθεώρηση του χρηματοοικονομικού κανονισμού θεωρούμε ότι αποτελεί μια καλή ευκαιρία προκειμένου να επικεντρωθούμε ακριβώς στα αποτελέσματα αυτά που επιθυμούμε. Η κυρία Λουμπαϊβά είπε ότι κατά τη διάρκεια του προϋπολογιτού της απαλλαγής καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή αντίληψη για το τι αποτελεί αποτελεσματικότητα και απόδοση. Αυτό είναι καλό σημείο κίνηση. Σε ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Και τώρα, τελευταία ερώτηση από την κυρία Αγιάλα Σέντερ. Αλλά σα παρακαλώ πολύ σύντομα, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ για την κατανόησή σα, κυρία Πρόεδρε. Απλώ γιατί πάντα είναι ενδιαφέροντα αυτά που μας λέει ο κύριος Λασάρου και θα ήθελα να του θέσω το εξή ερώτημα για τις ειδικέ εκθέσεις. Στο παρελθόν, σε κάποια στιγμή, η Επιτροπή μας είχαν την, είχε την εντύπωση ότι κάποιες από αυτές τις ειδικέ εκθέσεις επαναλαμβανόντουσαν, είχαν ένα χαρακτήρα επαναληπτικό για τα θέματα γεωργίας, διαλάμβαναν θέματα τα οποία ήταν κάπως πολύ ειδικά σε σχέση με τους γενικούς ε, στόχους κύριε Λαζάρου, ε, αν ανανεωθεί η θητεία σας και εξακολουθήσετε να έχετε κάποιες ε, αρμοδιότητες παράλληλες με τις προηγούμενες στο ελεκτικό συνέδριο, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να επιληθούν αυτά τα προβλήματα της επανάληψης ή της αλληλοεπικάλυψης για θέματα τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο περιορισμένες εμβέλειες Και επίσης πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα εθνικά, τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια να λύσουν τα προβλήματα που αναφέρατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γελασεντέρ. Μέσω της μεταρρύθμισης του Ελληνικού συνεδρίου για να προσανατολιστούμε στα αποτελέσματα και μέσω της νέας μεθόδου προγραμματισμού που ήδη εφαρμόζουμε δηλαδή η πρώτη μας προτεραιότητα να είναι ο σχεδιασμός που θα εγκρίνει βεβαίως το ελληνικό συνεδρίο, η κατανομή των ελέγχων, ανατμήματα και μετά βεβαίως όλα αυτά πρέπει να πάρουν τη μορφή ενός εγγράφου το οποίο θα συζητήσουμε στην ολομελία μας. Αυτό προϋποθέτει ορθή κατανομή των πόρων μας, ανά θέμα, ανά τομέα, Προποθέτει ότι θα είμαστε στην ώρα μας. Θα δημοσιεύουμε στοιχεία εγκαίρως για να μπορούμε να συμβαδίζουμε και με το δικό σας νομοθετικό έργο. Το πώς θα συνεργαστούμε καλύτερα είναι δική μας υπόθεση. Βεβαίως η συνθήκη φέρει το πλαίσιο μεταξύ του Ελληνικού Συνεδρίου και των χωρών μελών. Λέει δηλαδή ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε σε πνεύμα τη με ανεξαρτησία από την πλευρά μα και από εκεί πέρα έχουμε την Επιτροπή σα, την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και τις ομάδε εργασία. Εκεί εμεί πρέπει να εργαστούμε για να βρούμε νέους τρόπους δραστηριοποίησης για να γίνει η συνεργασία μας πιο αποτελεσματική. Η πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Λιζάρο και εγώ έχω κάποια, κάποια ερωτήματα, όμως με κάλυψαν οι προηγούμενοι και επειδή έχουμε καθυστερήσει θα δώσω τον λόγο στον Κεσόλτες, τον εισηγητή για, να, για μια κατακλείδα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λαζάρου για τις απαντήσεις του Θεωρώ ότι μας έδωσε πολύ επαγγελματικέ απαντήσεις και εγώ χάρηκα που κατέθεσε για άλλη μια φορά την πρόθεσή του να συνεργαστεί επικοδομητικά με την Επιτροπή μας και που μας επιβεβαίωσε ότι αργά αλλά σταθερά με πνεύμα ευθύνη στο ελληνικό συνέδριο θα προχωρήσει, θα βελτιωθεί εισακούγοντα και τις ανησυχίες και τα μελήματα και των άλλων εμπλεκομένων γιατί όλοι μας ε, εργαζόμεθα για το κοινό συμφέρον για να προστατεύσουμε τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χρήματα των φορολογουμένων, πατάσσοντας τις, τασταλίες, αλλά και φροντίζοντας να παρούμε τα χρήματα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ εκ μέρους της Επιτροπής μας για έξι χρόνια συνεργασίας, κύριε Λαζάρου. Ελπίζω ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ ένα λεπτό για να αποχωρήσει ο κ. Λαζάρου και να εισέλθει ο επόμενος υποψήφιος. Uh, Συνεχίζουμε με την μερική ανανέωση των μελών του Ελεκτικού Συνεδρίου. Καλώς ορίζω θερμά τον κύριο Λεμπρινκάτ, υποψηφίο εκ μέρους της Μάλτας. Χαίρομαστε που σας έχουμε εδώ σήμερα. Ξεκινούμε με την παρουσίαση από τον εισηγητή μας και εν συνεχεία ε, θα έχουμε την εισηγησία και ερωτήσεις από τα μέλη μας. Κύριε Σόλτος, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριος Σπρίγκατ, είναι γνωστός εδώ. Να αναφέρω απλώς λίγα πράγματα τα οποία νομίζω είναι σημαντικά. Ο ψήφιος είναι πολιτικός από τη δεκαετία του 80, πρόεδρος α, ε, της Επιτροπής Ελέγχου Εθνικών Λογαριασμών. Εργάστηκε την HSBC στην Μάλτα, Επίσης εργάστηκε για το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στο Λονδίνο. Επί δύο έτη ήταν υπουργό Οικονομικών και Εμπορίου και επί τρία έτη υπουργό Εφορικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Μεταβολής του Κλίματος. Περιμένουμε με ανυπομονησία την εισήγησή του. Ένα από τα επιτεύγματά του στο παρελθόν ήταν η συμβολή του στην σύσταση ενός εθνικού γραφείου ελέγχου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για κάθε χώρα. Ούτως ή άλλως υπάρχει ένα ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο δηλαδή, που θα ελέγχει τους εθνικούς λογαριασμούς. Ως υπουργό επίσης δημιούργησε μια ανεξάρτητη αρχή περιβάλλοντος και φυσικών πόρων ένα άνθρωπος που γνωρίζει τα του περιβάλλοντος, γνωρίζει και άλλα θέματα ε, ποιότητας. Ε. πολύ σημαντικά θέματα αυτά για κάθε χώρα. Κύριε Μπρινκάτ, παρακαλώ, πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Κύριε Μπρινκάτ, έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, γλυκτά μέλη της Επιτροπής, με αίσθημα Ευθύνη, έρχομαι εδώ ως υποψήφιο, εμφανίζουμε εδώ ως υποψήφιο της Μάλτας στο ελληνικό συνεδρίο έχω πίσω μου 30 χρόνια πείρα στον δημόσιο τομέα σε δραστηριότητε ε, που έχουν σχέση με τα χρηματοοικονομικά, την οικονομία, την δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς. Η ανεξαρτησία είναι βεβαίως κάτι απολύτως επιθυμητό. Αρχίζομαστε πείρα στην διαχείριση προγραμμάτων, σε έρευνες και σε υποβολή αναφορών και εκθέσεων. Η ανεξαρτησία όμως του ελεγκτή είναι η πιο σημαντική παράμετρος από την οποία εξαρτάται η αξιοπιστία κάθε ελέγχου. Είναι ο κρυγωνίος λήθος κάθε ελεγκτικής διαδικασίας. Το έχω δηλώσει απαντώντα το ερωτηματολόγιο ότι δεν πρόκειται να λάβω οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή από οποιοδήποτε άλλον φορέα και δεν πρόκειται να κάνω οτιδήποτε το οποίο δεν θα συναντεί 100% με τα καθήκοντά μου. Η έλεγχη του ελληνικού συνεδρίου και το γέννη έργο του πρέπει να είναι ποιοτικό και αξιόπιστο. Ο χρονισμός επίσης είναι πολύ σημαντικός γιατί πολλές φορές δύσκολα παρακολουθούμε εγκαίρως ε, διάφορες ευρωπαϊκές εξελίξεις. Πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπαθίες μας. Πρέπει να είμαστε ορατοί, να το προβάλλουμε το έργο μας, να είμαστε ευαίσθητοι, αλλά και αποτελεσματικοί σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά με απλούστερο τρόπο, με πιο αποδοτικό τρόπο, υποβάλλοντας εγκαίρως εκθέσεις, που θα εντοπίζουμε τα προβλήματα. Πρέπει επίσης οι ελεγχόμενοι να βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν τις συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου, κατά τη γνώμη μου, είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να λάβουμε πρωτοβουλίες επικοινωνιακές προς τους πολίτες μας, που είναι και οι τελικοί δικαιούχοι, οι τελικοί ωφελούμενοι από τις ε, ακαμπτές προσπαθίες μας, να βελτιώσουμε και το έργο μας, αλλά και στο πλαίσιο του τονισμού ότι το έργο μας είναι ενιαίο. Ποιότητα, αξιοπιστία είναι βασικές μας ε, αρχές. Επίσης, το έργο μας δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό, είναι διαρκές και αυτό πρέπει να γίνει συνειδητό. Ε, εάν ε, επιδοθεί ο διορισμός μου, εγώ προσωπικώς θα δράσω και θα αναλάβω πρωτοβουλίες έτσι ώστε οι εκθέσεις μας πέρα από τα γενικά θα αποτελέσουν και πιο συγκεκριμένα βάση για περαιτέρω ενεργική διαβούλευση και διάλογο με τους διάφορους εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των πολιτών. Όλα αυτά θα διευκολύνουν τη διαδικασία που όλοι επιθυμούμε για περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη απόδοση, λογοδοσία και ευελιξία. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς ελέγχου και εγγυήσει σε διαθεσμικό επίπεδο, τόσο εντό όσο και εκτό του ελεγκτικού συνεδρίου. Στο πνεύμα ενισχυμένη συνεργασία πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο κοντά, να υπάρχουν περισσότεροι δεσμοί και φορεί επικοινωνία μεταξύ των δύο οργάνων. Ιδιαίτερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Οι επαγγελματικέ μου δραστηριότητε ήταν ανέκαθεν υπέρ τη καλή διακυβέρνηση της ε, διαφάνειας όσον αφορά τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά και όπως ήδη είπαμε ε, έχω υπηρετήσει στο Εθνικό Ελληνικό Συνεδρίο και δημιούργησε την πρώτη, το πρώτο ανεξάρτητο γραφείο δημοσιονομικού ελέγχου στη Μάλτα. Ήμουν ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος ε, επίσης της Επιτροπής Κρατικών Λογαριασμών. Τα παρακολούθησα αυτά από πολύ κοντά, όχι μόνο στην Μάλτα αλλά και στο εξωτερικό. Έχω υπηρετήσει σε διάφορες υπουργικέ ε, θέσεις, γνωρίζω και το νομοθετικό έργο, αλλά και τον δημοσιονομικό σχεδιασμό, τη διαδικασία κατάρτιση του προπολισμού κλπ. Καθώς και τις αρχές της καλής δημοσιονομικής διακυβέρνησης και εποπτείας. Έχω λοιπόν υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις που έχουν πάντα σχέση με την οικονομία και τα δημοσιονομικά. Αυτά ήταν ε, ανέκαθεν στο προσκήνιο κάθε φορά που χειριζόμουν και άλλα θέματα όπως την COP21 για το περιβάλλον ή στην θέσπιση εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το κλίμα στην Μάλτα. Αυτή ήταν και η πρώτη στρατηγική στη Μάλτα η οποία έθεσε την εφορία στο προσκήνιο. Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου, από την πλευρά μου θα συμβάλλω στην ενίσχυση του ελεγκτικού συνεδρίου ως εξωτερικός ελεγκτής. Πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη συνέχεια η απόδοση των ελέγχων να παραμείνει προτεραιότητα και για τους τρεις τύπους ελέγχου που διενεργεί το ελεγκτικό συνέδριο. Οι καθυστερήσεις πρέπει λοιπόν να μειωθούν, να εξορθολογήσουμε τη χρήση, την αξιοποίηση των πόρων μας και να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε. Πρέπει να συμμετέχουμε περισσότερο στον έλεγχο των κοινωτικών δαπανών, να βελτιώσουμε τη μέθοδο των ελέγχων, να πλουστεύσουμε τους μηχανισμούς και να ενημερώσουμε, να εξυγχρονίσουμε τους κανόνες μας. Και όλα αυτά ε, πρέπει να γίνουν γνωστά ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι, όχι μόνο για την αξιοποίηση των κοινωτικών πόρων, ε, αλλά και σε κάθε άλλη τομέα. Στο τομέα τη συμμόρφωση, ε, στο τομέα τη άμεση ή επιμερισμένη διαχείριση. Και τη άμεση και τη επιμερισμένη διαχείριση. Επίση, έχω την άποψη ότι ο προπολισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα τι στρατηγικέ μα προτεραιότητε. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσει, αλλά και ευελιξία. Το μέσω πρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίση, χρειάζεται και αυτό αναθεώρηση για να ενσωματώσουμε, όπω είπε τι προτεραιότητέ μα και χρειάζεται μια νέα ορμητικότητα για περισσότερη εποπτεία. Χρειάζεται επίση οι μηχανισμοί έγκριση των δαπανών να είναι πιο ευέλικτοι και είναι πλέον καιρό να αυξήσουμε την προστιμένη αξία μα, να σταλάξουμε ένα νέο πνεύμα δυναμισμού, να γίνουμε πιο δραστήριοι σε ένα συνεχώ μεταβαλλόμενο κλίμα στο ηλεκτρικό συνέδριο. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμεθα σκληρά σε όλα τα επίπεδα λοιπόν, του έργου μας. Να είμαστε να επαγρυπνούμε όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων και την αξιοπιστία τους κάθε φορά, τα οποία λαμβάνουμε εγκαίρως, ε, ελπίζουμε, από τους ενδιαμέσους. Χρειάζεται επίσης ε, να σημειωθεί πρόοδος στις επαφές μας με την ε, Επιτροπή και τα άλλα ελεγκτικά όργανα, αλλά και εντός του ελληνικού συνέδριου. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τις υφισταμένες ρυθμίσεις, γιατί αυτό θα μας κάνει πιο αποτελεσματικού στις επαφές μας με την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε μεγαλύτερη ελεπίδραση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. 80% των ε, κοινοτικών πόρων είναι αντικείμενο επιμερισμένη διαχείριση. Χρειάζεται να βελτιώσουμε την ποιότητα αυτή τη διαχείριση, χωρί βεβαίω να, εμπλακούμε άμεσα στη διαχείριση και του τελευταίου ευρώ. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε το έργο μα πιο γνωστό, να επικοινωνήσουμε καλύτερα, όντα πιο κοντά, όσο πιο κοντά γίνεται στου πολίτε μα. Διασφαλίζοντα ότι βεβαίω και το ελληνικό συνέδριο έχει τα ωριά του. Μπορούμε όμω να νομοθετήσουμε καλύτερου κανόνε. Αυτή είναι η ευθύνη μα η οικονομική ευθύνη, η ευθύνη τη οικονομική διακυβέρνηση. Το ελληνικό συνέδριο θα ενισχύσει κατόπιν όλων αυτών και τον δικό του ρόλο, το ίδιο το ελληνικό συνέδριο, αλλά και του άλλου εμπλεκομένου. Αν αποτύχουμε, αυτό θα υπονομεύσει τον διαλόγο ύπαρξη του ελληνικού συνεδρίου. Αν πετύχουμε όμω, θα ενισχύσουμε και την δημοκρατική ευθύνη ελέγχου που έχει το Ελληνικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε που παρουσιάσατε το έργο σας και θα κάνουμε κάποιες επιπρόσθετες ερωτήσεις. Ε, καταρχάς έχουμε τον εισηγητή μας, την κ. Σόλτα, ο οποίος θα θέσει ερωτήματα. Α, προτιμάτε να κλείσετε το γύρο των ερωτήσεων, μάλιστα. Ο κύριος Σαραβέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα προσωπικά σχόλια αυτά που κάνατε κύριε Μπρίνκατ. Θα καταλαβαίνετε βέβαια ότι ενώπιον της Επιτροπής μας θα πρέπει να τηρούμε τα πιο υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά τον διορισμό μελών του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Το Ελεκτικό Συνέδριο δεν αποτελεί ένα οποιοδήποτε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φήμη και το κύρος του θα πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητα και πέραν κάθε αμφιβολίας. Οποιοδήποτε ε, αμφιβολία για την ανεξαρτησία του λεκτικού συνεδρίου θα έβλαπτε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον αυτό θεωρώ εγώ. Δύο ερωτήσει, λοιπόν έχω να σας κάνω. Στην ε, πρόσφατη, στις πρόσφατες απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις που σας αποστήλαμε για το πώς αντιμετωπίζετε την ε, διαφθορά σε ό,τι αφορά τα άτομα από την χώρα σας, απαντήσατε με μεγάλο βαθμό λεπτομερίας και μας διαβεβαιώσατε ότι θα εξασφαλίζετε ότι το δικαστήριο, το ελληνικό συνεδρίο, συγγνώμη, θα διεξήγαγε πλήρη έρευνα όχι μόνο για να διορθώσει τυχόν ε, παραπτώματα, αλλά και προληπτικά. Ως ε, υπουργό στη Μάλτα, ένα από τα μέλη της ε, κυβέρνησής σας ε, είχε έκθεση στην υπόθεση με τα έγγραφα του Παναμά. Και ψηφίσατε στη συνέχεια να παραμείνει στην κυβέρνηση και έκτοτε αρνήσετε πεισματικά να σχολιάσετε το γεγονός αυτό. Και μια και είναι ο μοναδικό υπουργό τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματικά είχε εμπλοκή στην υπόθεση με τα έγγραφα του Παναμά, θα πρέπει να ξέρουμε το αν μπορούμε να εμπιστευτούμε και πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί τι θα γίνει άμα ξαναπροσδιοριστεί μια τέτοια περίπτωση και μάλιστα με το ίδιο άτομο ενδεχομένω στο ιστορικό της Ένωσης. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα αντιδρούσατε με τον ίδιο τρόπο αν είσαστε μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Πώς μπορεί να είμαστε σίγουροι. Και κατά δεύτερον, είπατε ότι ανεξάρτητα από τη δική μας άποψη της Επιτροπής μας δηλαδή και της Ολομέλειας θα συνεχίσετε να είστε υποψήφιος ανεξάρτητα από την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Άρα το ερώτημά μας είναι απλό. Προτίθεστε να δεσμευτείτε τώρα ενώπιόν μας ότι θα σεβαστείτε την απόφαση της Επιτροπής και αν υπήρχε κάποια διαφορετική τοποθέτηση, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα θα σεβόσαστε την άποψη του Κοινοβουλίου, όπως θα την εκφράσει η Ολομέλεια. Μάλιστα, κύριε Μπρίνκατ, έχει το λόγο για να απαντήσει. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω, αγαπητές συνάδελφοι από τη Φιλανδία, και να ξεκινήσω με τη δεύτερη ερώτηση, σε ό,τι αφορά την ερώτηση υπαριθμό 19. Πέραν από αυτά που είπα λοιπόν στο ερωτηματολόγιο, με ρωτάτε, αν σωστά σας καταλαβαίνω και διορθώστε με αν κάνω κάτι λάθος, αν σέβομαι τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Ναι, θα σεβαστώ αυτά που θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο και προφανώς θα αφήσω τα πράγματα αυτά στα δικά σας χέρια να με αξιολογήσετε βάσει δύο ζητημάτων όμως των ικανοτήτων μου και της ακυριότητάς μου. Και αυτό με φέρνει ε, στο πρώτο ερώτημα που θέσατε σε ό,τι αφορά τα έγγραφα του Παναμά και την ε, ψηφοφορία που έγινε στο Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν 36-41 οι ψήφοι οι οποίοι ε, είχαμε τότε στο Κοινοβούλιο. Άρα δεν ήταν δική μου η ψήφο η καθοριστική. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερον, έχω εδώ ένα έγγραφο με ημερομηνία 20 Απριλίου και επικεφαλίδα Ελευθερία ελευθερίας ε, ψήφου σε ό,τι αφορά τα θέματα ψηφοφορία στο Κοινοβουλίο αυτό. Και όπως είπατε, αυτό το θέμα δεν είναι τόσο θέμα συζήτησης, όσο θέμα συνείδησης ε, στη Μάλτα. Όπως ε, επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από έναν συνταγματιολόγο, έχουμε το σύστημα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, το οποίο ουσιαστικά τι προκαθορίζει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες οποιοδήποτε παραβιάζει α, τη γραμμή την κυβερνητική ή του κόμματος μπορεί είτε να αποβληθεί είτε να ατυχθεί από την κοινοβουλευτική του ομάδα, από το κόμμα του. Για να σας το πω αξιπτοδοτία δεν είχα επιλογή. Δεν είχα επιλογή, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω και το εξής. γιατί αν ε, καταλάβατε σωστά Είπατε ότι δεν το σχολίασα το ζήτημα αυτό ποτέ εκ των υστέρων. Εδώ έχω μία αντίρρηση, γιατί έχω διάφορες δηλώσεις να σας υποβάλω για διάφορες κατηγορηματικές δηλώσεις μάλιστα στις οποίες ε, προέβηκα. 22 Μαρτίου του φετινού έτους στη Μάλτα ανέφερα ότι αν γίνει το σφάλμα αυτό η κυβέρνησή μου, γιατί τότε ήμουν ε, υπουργό. η κυβέρνησή μου λοιπόν ε, διακινδυνεύει να υπονομεύσει την ίδια της την επιτυχία. Και τότε λοιπόν ξεκαθάρισα τότε ότι πρόκειται για το δεύτερο κυβερνητικό στέλεχος ε, που έκανε σχετικέ δηλώσει για τα έγγραφα του Παναμά. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ λοιπόν ότι μίλησα και ανέφερα ποια ήταν η άποψή μου μίλησα για πραγματική υπονόμευση τη επιτυχία τη κυβέρνηση. Και κάτι άλλο θα ήθελα να δείξω, το οποίο δεν το δείξατε εσεί, αλλά πιστεύω ότι είναι σχετικό. Μήπω θα έπρεπε να έχω εξετάσει το ενδεχόμενο να παρατηθώ. Το εξέτασα. Και αυτό που επικράτησε ω σκέψη ήταν το εξή, ότι εάν παρετούμουν στο Μαλτάζικο Κοινοβούλιο τουλάχιστον, για μία ημέρα θα ήμουν ο ήρωας. Αλλά στην τελική ανάλυση δεν θα ακουγόταν πουθενά αλλού η φωνή μου. Ειλικρινά πιστεύω ότι συνεχίζοντα τι εργασίε μου στα πλαίσια των δομών αυτών, όσο περνισμένη και αν είναι η σύμβολή μου, εξακολουθώ να αποτελώ μία α, φωνή η οποία μιλά και προ μία άλλη κατεύθυνση. Και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο δεν παρατήθηκα. Όταν έγραψα όμω το άρθρο αυτό εδώ πέρα, ήταν πριν ε, την ψηφοφορία. Και επανέλαβα τις απόψεις μου αυτές και μετά την ψηφοφορία και εξακολουθώ να υποστηρίζω λοιπόν την άποψη αυτή. Και μάλιστα έγραψα και ένα σχετικό άρθρο στα Μαλτέζικα με τίτλο «Θα πρέπει να αποτελέσουμε πηγή έμπνευσης» γιατί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργό μας μας είχε, πει, είχε δηλώσει ότι θα πρέπει να αποτελούμε πηγή έμπνευση και φιλοδοξία για την κοινωνία. Και εγώ προσέθεσα το εξή και διευκρίνησα το εξή ότι ναι, να είμαστε πηγή έμπνευση, αλλά να δώσουμε και στον κόσμο την ε, εντύπωση και την ελπίδα ότι δίνουμε εξίσου μεγάλη προσοχή σε θέματα Κοινωνική ανάπτυξης και δικαιοσύνη, όπως και στα θέματα οικονομικής ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν έτσι απάντησα στι ερωτήσει σα. Ναι, μια διευκρίνηση. Μία πρόταση μόνο. Αν ο ίδιο υπουργό, αν εσείς είσαστε μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου και καλούσασταν να αποφασίσετε για τέτοια ζητήματα, Ω μέλο του Ελληνικού Συνεδρίου, θα αισθανόσαστε ότι έχετε την ελευθερία να εκφράσετε τι απόψει σα και να δράσετε αναλόγω. Ω ουδέτερο μέλο. Ναι, θα πήγαινε και ένα βήμα παραπάνω. Ακόμα και αν δεν ήμουν μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, να σας πω ότι θα έκανα δύο ενακτικές, θα εξέταζα είτε να παρατηθώ, είτε να βγω από την κοινοβουλευτική ομάδα και από την κυβέρνηση μέχρι να καθαριστεί το όνομά μου, όχι μόνο από νομική άποψη, γιατί να είμαι ειλικρινή, δεν είμαι βέβαιο ότι υπήρξε παράβαση νόμου, αλλά από δεοντολογική άποψη. Όπω είχε πει και ο πρόεδρο Ομπάμα, υπάρχουν τα νομικά ζητήματα, αλλά υπάρχουν και τα δεοντολογικά ζητήματα. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα πρόσωπο με ένα άτομο με πολιτική έκθεση, υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά τα θέματα νομιμότητα και δεοντολογία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρίνκατ. Έχω την κυρία Ίνες Αγιάλα Σέντερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Κύριε Μπρινκάτ, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και τις εκτενείς απαντήσεις που έχετε δώσει. Και εγώ για να διαλυθούν οι παρεξηγήσεις θα ήθελα να πω στον κύριο Σαβαρμά κ. Ματέας δεν είναι ο μόνος ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Ο κ. Σόρια, ο Ισπανός υπουργό ε, Βιομηχανίας, είναι το πρώτο άτομο το οποίο φαίνεται να εμπλέκεται στα έγγραφα του Παναμά. Δεν ε, παρετήθηκε, είπε ψέματα ότι δεν είχε καμία σχέση και μετά αναγκάστηκε να το παραδεχτεί και μετά φυσικά αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Υπάρχουν και άλλοι υπουργοί που φαίνεται ότι εμπλεκόντουσαν αλλά δεν θέλησαν να εξέλθουν από την κυβέρνηση. Προφανώς εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω μια τέτοια στάση και δεν, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για το θέμα της Μάλτας, αλλά ξέρω ότι εσείς ε, ήδη για να γίνετε υποψήφιος για το ελεκτικό συνέδριο παραιτηθήκατε από το υπουργικό αξίωμα. Είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι περιμένουν να δουν αν θα εγκριθούν και εάν όχι παραμένουν οι υπουργοί. Εσεί τουλάχιστον παρατηθήκατε από το αξίωμα του Υπουργού για να γίνετε υποψήφιο για το ελεκτικό συνέδριο, κάτι το οποίο μου φαίνεται ότι ήταν μια σημαντική ενέργεια. Αναγνωρίζω επίση ότι το έργο που έχει γίνει από τη Μάλτα, που είναι μια χώρα του Νότου, όπου το θέμα του περιβάλλοντος είναι πάντα πιο ευαίσθητο και πιο δύσκολο να εφαρμοστεί ακριβώς λόγω των κλιματικών περιορισμών και πιέσεων που υπάρχουν, νομίζω ότι ο ρόλος σας ήταν πάρα πολύ σημαντικός ως εκπροσώπου της Μάλτας για να μπορέσετε να πιέσετε για μια τελική συμφωνία στην COP21. Εμείς ως Ευρώπη τώρα αυτή τη στιγμή υπολοιπόμεθα άλλων χωρών στον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα εσείς κάνατε μια μεγάλη προσπάθεια. Εδώ, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω <clears throat> είναι σε σχέση με την εμπειρία σας. Είπατε ότι είχε εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, στον τραπεζικό τομέα και φυσικά έχουμε μεγάλα προβλήματα στα θέματα αυτά γιατί το ελεκτικό συνέδριο αρχίζει πραγματικά να ασχολείται με το τμήμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που είχε να κάνει με την επίλυση των τραπεζικών προβλημάτων των κρατών μελών, τις κρατικές εγγυήσεις και τα λοιπά που εδόθηκαν και θα ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς από τη δική σας οπτική γωνία και με την εμπειρία σας πώς βλέπετε αυτή την ανάγκη να υπάρξει πραγματικά έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μέσα σε διάφορα εργαλεία μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μέσω των ιδιωτικών τραπεζών χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν αυτά τα κονδύλια. Και επίσης επί τη βάση της εμπειρίας σας για τη δημιουργία του πρώτου εθνικού οργανισμού στη Μάλτα για ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο, με ποιο τρόπο βλέπετε την δυνατότητα αυτή να προωθηθεί, να ενισχυθεί η δυνατότητα των εθνικών ελεκτικών συνεδρίων που σε πολλές χώρες περίπου με δυσκολία κινούνται και δρούν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κράτη τα συνεδρία αναγκάζοντας τα κράτη-μέλη να είναι πιο διάφανα στον τρόπο που εφαρμόσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έρχεστε από μια πιο μικρή χώρα από τη δική μου, που δεν έχει τόσο μεγάλα προβλήματα βεβαίω όσο η δική μου, αλλά παρόλα αυτά τα δικά σας προβλήματα μπορούν να μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και η άποψη που έχετε για το πώς μπορούν να επιληθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρίνκατ. Κυρία Σέντερ, τρία κύρια ερωτήματα πιστεύω ότι μου θέσατε. Για το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι πάντα πρόκληση, ιδίω σε ένα μικρό νησί όπως η Μάλτα που έχει περιορισμένη έκταση, μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού και τα προβλήματα που έχουν τα νησιά της Μεσογείου. Παράλληλα όμως να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι ότου ανέλαβα τα καθήκοντά μου, το περιβάλλον στην Μάλτα δεν είχε κάποιο καν ρυθμιστικό φορέα. Ήταν τμήμα ενός φορέα, μιας αρχής που λεγόταν ΝΕΠΑ και η οποία ουσιαστικά ήταν προσανατολισμένη στην χωροταξική σχεδίαση. Και όταν εμείς εξελέγημε, όταν η κυβέρνηση στην οποία μετήχα εξελέγει, θέλησαμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον περιβαλλοντικό φορέα με ανθρώπους, κύρους, αξιο, και υψηλού πολιτικού προφίλ. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο έχει γραφεί, υπάρχουν πολλά θα πω γραφεί μάλλον από μέλη του Κοινοβουλίου της Μάρτας που επενούν την σύνθεση αυτής της ανεξάρτητης αρχής για το περιβάλλον. Όταν του συνάντησα λοιπόν μαζί με τους ε, εργαζόμενους, εκπρόσωπους εργαζομένων και μαζί με τη, το Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ θέλησα να δώσω δύο σημαντικά μηνύματα. Τους είπα ότι δεν θα παρέμβω στην καθημερινή διαχείριση του φορέα Μόνο αν κάποιος πιο ψηλά προσπαθήσει να παρέμβει στις δραστηριότητές της, δραστηριότητές σας για να τον αποτρέψω και του είπα επίσης ότι έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Πρέπει να είσαστε, πρέπει να είσαστε οι φύλακες να παρακολουθείτε και να προστατεύετε τα θέματα του περιβάλλοντος. Τώρα, όταν παρετήθηκα, λόγω της τρέχουσας υποψηφιότητας, είχε μόλις δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, μια σειρά αποδομές, για να προχωρήσει αυτή η αρχή και είχαν καθοριστεί τα καθήκοντά τη και ήταν στη φάση τη δημιουργία ικανοτήτων. Δεν μπορώ να, να λοιπόν την ευθύνη για αυτά που έγιναν πέραν του Μαΐου εφέτο, αλλά είμαι υπερήφανο και πιστεύω ότι είναι πολλέ από τι αποφάσει που ελήφθησαν στη Μάλτα που δεν θα ήταν δυνατέ χωρί την ύπαρξη αυτή τη περιφαλλοντική αρχή. Γιατί αλλιώ ήταν μια ε, γενική διεύθυνση μέσα σε μια αρχή η οποία είχε να κάνει με τα θέματα σχεδιασμού. Για τον τραπεζικό τομέα και τη σχέση μου. Ε, τη στιγμή αυτή που υπάρχουν πολλές τράπεζες οι οποίες είναι κάτω από τα φώτα της επιχειρότητας, όπως παραδείγματος για τα σκάνδαλα LuxLeaks και τα έγγραφα του Παναμά, οι τράπεζες στις οποίες εργάστηκα πάντα ήμουν εκεί ως ένας ε, διαχειριστής σε υψηλό επίπεδο. Δεν υπήρξα ποτέ διεθνός σύμβουλος, δεν υπήρξα μέτοχος δεν είχα εμπλακεί επομένως ποτέ στη διαμόρφωση πολιτικής. Και τα τελευταία χρόνια που ήμουνα στο τραπεζικό τομέα ήμουνα αρμόδιος για τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής, δηλαδή έρευνα σε σχέση με διάφορες υπηρεσίες της τράπεζας αυτής. Για να απαντήσω και στο ερώτημα σας λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τροποποίηση, μια μεταρρύθμιση στον τραπεζικό τομέα μετά από τα σκάνδαλα LuxLeaks και του Παναμά. Πρέπει κανείς λοιπόν να δει αυτόν τον τομέα ο οποίος αλλάζει με ένα πάρα πολύ δυναμικό τρόπο. Η Μάλτα έχει ξεπεράσει την, το τραπεζικό απόρριτο πολύ πιο πριν από άλλες χώρες στην Ευρώπη και στην ε, Μάλτα με τις πληροφορίες που έχω είναι ότι η Μάλτα πάντα συμμορφώθηκε στο τραπεζικό τομέα και στα θέματα απορρίτου και τα λοιπά με τα, και τη διαφάνεια με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Άλλη έχει σειρά να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπρινκάτ, κατά πρώτον την εξαιρετική εισήγησή σας είναι εξίσου εντυπωσιακό και το βιογραφικό σας. Έχετε τόση πείρα. Αυτό χρειαζόμαστε και στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς, να εκλέξουμε κάποιον ο οποίος θα τα καταφέρει. Και εκτίμησα και την πρότασή σας υπέρ της απλούστευσης των ελεγκτικών διαδικασιών. Ε, ξέρετε, είναι η δεύτερη θητεία μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρώτη φορά του. Έχω περάσει από τότε, ξέρω, 10 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ε, θυμάμαι ότι και από τότε μιλούσαμε για απλούστευση. Και δυστυχώς από τότε, μετά από 10 χρόνια, βρισκόμαστε στο, πάλι στην αρχή. Τίποτα δεν έχει γίνει. Ελπίζω πάντως ότι αν ξεκινήσουμε έστω και από το ελληνικό εκτικό συνέδριο, καλό θα ήταν. Να ξεκινήσουμε από κάπου. Εσείς πώς το βλέπετε, πώς βλέπετε να ξεκινάει αυτή η απλούστευση. Ας ξεκινήσουμε από τις εκθέσεις, θα ήταν καλό. Αλλά θα μπορούσε και η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διευθύνσεις να κάνουν το ίδιο. Και θα έπρεπε μάλιστα. Και δύο ακόμη ερωτήσεις με απόδοση και αποδοτικότητα. Μιλούμε για την πράσινη ανάπτυξη. Το έχετε εφαρμόσει ποτέ. Για την επίτευξη προσθέμενης αξίας και το άλλο αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα τον οποίο έχετε υπηρετήσει. επιμείνετε από ό,τι άκουσα στην αποδοτική διαχείριση πόρων και ελέγχων και Ξέρω ότι θέσετε στόχους στον προϋπολογισμό και τους στόχους αυτούς τους μεταφράσετε σε ποσοτικούς στόχους. Υπάρχουν τέτοιοι στόχοι, που δεν πετύχατε ή που θα θέλετε να αναθεωρήσετε και πώς θα μεταφράσετε τους γενικότερους στόχους σε ποσοτικούς στόχους και ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί εξ αυτών κατά τη γνώμη σας η απλούστευση είναι πολύ σημαντική. Χωρίς απλούστευση θα υπάρχουν επικαλύψεις, θα έχουμε χαμηλότερη απόδοση, θα έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία και θα λέγω ότι θα δημιουργούσαμε και χώρο για διαφθορά. Αυτά ισχύουν για κάθε χώρα και για κάθε θεσμικό όργανο. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε απλούστευση. Το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να αλλάξει εσωτερικά, όπως και όλα τα άλλα θεσμικά όργανα, άλλωστε. Ας δούμε τον ε, κοινωτικό προπολισμό. Πρέπει να προσαρμοστεί στις στρατηγικές ανάγκες. Πρέπει η νομοθεσία να γίνει πιο αποτελεσματική, να εξορθολογιστεί. Πρέπει να διευρύνουμε επίση την εντολή μας. Και το λέω εξωτερικός αυτή, ακόμη, το ελεγκτικό συνέδριο ορθώς από τον καθαρά οικονομικό έλεγχο περνάει στην οικονομική διακυβέρνηση. Υπάρχει αυτή η μετακίνηση, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους τους εμπλεκομένους. Όμως το πιο σημαντικό είναι να μην περιοριστούμε στη διατύπωση εκθέσεων. Το να γράφουμε εκθέσεις είναι ένα. Το να υλοποιούνται είναι το πιο σημαντικό. Οι συστάσει λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, με σοβαρότητα και αυτό θα μας κάνει πιο αποτελεσματικούς στην εφαρμογή. Ακόμα και οι ειδικέ εκθέσεις, εξαιρετικά αξιόλογες, πρέπει να διατυπώνονται, θα έλεγα, απλούστερα, ταχύτερα, έγκαιρα. Το χρειάζεται αυτό το ελληνικό συνέδριο, πρέπει να επανεφεύρει τον εαυτό του. Επίσης χρειαζόμαστε περισσότερες περιοδικές τακτικές συναντήσεις με τα κρατημέλη. Θεωρώ ότι δεν είναι επαρκής η σημερινή ίσως και σε συνεργασία και σε επαφή με τα εθνικά γραφεία ελέγχου. Ίσως κάποια έλεγχη πρέπει να γίνονται συνεργατικά, σε, ανάλογα με το επίπεδο φυσικά με το κράτο μέλο. Και βεβαίω να περιορίσουμε τι επικαλύψει των ελληνικών εργασιών. Δεν ξέρω αν απέντησα σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ε, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θίξω κατά κλείδι. Παλιά όλοι είχαμε στόχο την απορρόφηση. Σήμερα ξέρουμε ότι το να απορροφάς απλώς πόρους δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε αποτελέσματα. Πρέπει οι πόροι να δαπανώνται για να βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών. Και βεβαίως περισσότερη η λογοδοσία από την πρώτη στιγμή, τη διάθεση των πόρων, ως την επίτευξη των αποτελεσμάτων, την εκτέλεση των εργασιών. Πρέπει να βλέπουμε απτά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση. Και να φύγουμε από την νοοτροπία του να ξοδέψουμε ό,τι έχουμε. Όχι απορρόφηση αλλά μέσω εξορθολογισμένης επένδυσης σε πραγματικούς στόχους. Να επενδύουμε λοιπόν στην επίτευξη των στόχων του 2020. Αυτά είχα να πω. Αν ξέχασα κάτι παρακαλώ ε, να μου το επισημάνετε. Ευχαριστώ. Λέει πρόεδρος. Ήμουν και εγώ στον καταλόγο των ομιλητών. Τρεις ερωτήσεις, νομίζω εύκολες και σύντομες. Πρώτον, αν καταλάβα καλά, ότι το γραφείο ελέγχου στην, Άλτα, στη Μάλτα. Είναι, είναι γραφείο της Βουλής. Ε, πώς ε, διασφαλίζεται η εξαρτησία αυτού του γραφείου της Βουλής. Επίσης αναφέρεται κατά παράληψη τον όρο καλή διακυβέρνηση, συνοχή, δημόσια λογοδοσία κλπ. Που είναι και ο στόχος της ε, Επιτροπής μας Ελέγχου του Προπολισμού και του Ελεγκτικού Συνεδρίου φυσικά. Τη διαφάνεια τη λαμβάνουμε πολύ ε, υπόψη μας στα σοβαρά. Η κυβέρνηση στην Μάλτα της οποίας ήταν μέλος ε, επικρίθηκε στα μέσα λόγω του ότι δεν ε, κατάφερε να δημοσιεύσει στοιχεία σχετικά με δημοσίες προμήθειες, δημοσίες συμβάσεις, ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα. Δεσμεύεστε να βελτιώσετε τη διαφάνεια ως ε, μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου και τι συμβουλή θα δίνετε στα άλλα κράτη-μέλη ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Και τρίτον, επιτρέψτε μου, μια πολύ προσωπική ερώτηση. Τουλάχιστον έτσι τη βλέπω εγώ, γιατί το 2004, όταν εμεί ε, και οι χώρε μα, δηλαδή και οι δύο χώρε μα, ήταν μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ ήμουν ε, υπέρ τη ένταξη τη ε, Τσεχία, την υποστήριξα θερμά. Και δύσκολα θα άλλαζα γνώμη. Οπότε θέλω να σα ρωτήσω πώ άλλαξε η γνώμη σας μετά από την ένταξη της Μάλτας. Είναι μια, έτσι, θέλετε, προσωπική περιέργεια, αλλά είναι σημαντική επάντηση για μένα. Σας ευχαριστώ για τις τρεις αυτές ερωτήσεις, πολύ ε, επίκαιρες. Καταρχάς να σας εξηγήσω τι ήταν και τι είναι σήμερα, τι ήταν στο παρελθόν και τι είναι σήμερα αυτό το ελεκτικό συνέδριο στη Μάλτα. Στις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν παράρτημα του Υπουργείου Οικονομικών. Έμεσα ή έμεσα ή άμεσα ήταν υπό την επιρροή του Υπουργού. Άρα δεν είχε οποιαδήποτε αυτονομία και ανεξαρτησία. Και η προηγούμενη η κυβέρνηση και η δική μου κυβέρνηση όμως το 1996 δεσμεύτηκαν να εγγυηθούν πραγματικά την ανεξαρτησία ε, της υπηρεσίας αυτής. Και το 1997 λοιπόν ε, με σχετική νομοθεσία και υποστήριξη και των δύο κομμάτων ε, άλλαξαν τα πράγματα και άρα σε κάθε περίσταση ο Γενικός Ελεγκτής ήταν, διοριζόταν μετά από συνένεση και των δύο κομμάτων και των δύο πλευρών. Σήμερα τώρα, η ηλεκτρική υπηρεσία αυτή α, ενεργά εντελώ ανεξάρτητα και ποτέ δεν υπήρξε οποιαδήποτε υποψία από προηγούμενη τρέχουσα ή μελλοντική κυβέρνηση. Κανεί λοιπόν στη Μάλτα, εκτό ίσω από το κόμμα τη Εκκλησία που ενδεχομένω να διαφωνεί με τα πορίσματα της Επιτροπής, δεν έχει αμφισβητήσει τη λειτουργία της. Αυτό το τονίζω. Είναι πραγματικά υψηλά το κύριο στο οποίο απολαμβάνει αυτό το σώμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, δημόσιες συμβάσεις, ε, σωστό το ερώτημα. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να υπάρχει εμπιστευτικός χαρακτήρας. Και ξέρω ότι τα πράγματα είναι ε, πολύ ευαίσθητα. Όταν υπάρχουν ε, όμως ε, μεγάλες συμβάσεις, είναι προς το όφελος του κοινού να δημοσιεύονται τα έγγραφα αυτά για δύο λόγους. Όχι μόνο για δημόσια κατανάλωση, αλλά γιατί. Ως αποτέλεσμα της Επιτροπής Δημοσίων Λογαριασμών και ήμουν συνειδητρητής της Επιτροπής αυτής, ε, έχω να σας πω το εξή ότι όταν δημοσιεύονται αυτές οι επαφές μπορούν να περάσουν πλήρη έλεγχο της σχετικής επιτροπής ε, του Κοινοβουλίου και της υποεπιτροπής μέχρι ότου δημοσιευτούν όμως δεν μπορούν να ελέγχονται. Δεν μπορεί να ελέγχονται συμβάσει που δεν έχουν δημοσιευτεί, άρα πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τίθεται μια τέτοια καταρακτική ημερομηνία από την ε, κυβέρνηση και να τηρείται αυτή η προθεσμία. προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία ελέγχου των συμβάσεων αυτών. Και φυσικά υπήρξαν και συμβάσει στο παρελθόν ε, πολύ ευαίσθητε, για παράδειγμα για την παραγωγή πετρελαίου κτλ. Ε, οι οποίε πέρασαν από αυστηρό έλεγχο και παρόλα αυτά υπήρχαν ζητήματα. Και τέλο, να περάσω στο τελευταίο ερώτημα. Ποτέ δεν ήμουν κατά τη Ευρώπη. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ποτέ σε καμία περίπτωση, αντίθετα με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αντιθέτως, είχαμε πει ότι αν ο κόσμος αποφασίσει μέσω των γενικών εκλογών ότι θέλει η χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το κόμμα μου θα άλλαζε άμεσα τοποθετηθεί. Και αυτό συνέβη. Και μάλιστα μέσω των δράσεων του κόμματος μου, όχι μέσω των στρατηγικών δηλώσεων. Άρα, ενεργά συμμετείχα στα πλαίσια και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσουν πολλοί μεταξύ των οποίων και ο συνάδελφο ε, ο κ. Τζάξον τη αντιπολίτευση, γιατί συνεργαστήκαμε στενά για να προωθήσουμε λοιπόν τι ιδέε και την τοποθέτηση τη ε, Μάλτα στα διεθνή φόρα. Και σε τα πλαίσια διαφόρων ε, θεσμικών οργάνων, λοιπόν, έχω προασπίσει τα συμφέροντα αυτά. Και να σας πω ότι ως Υπουργός Περιβάλλοντος δραστηριοποιήθηκα ιδιαιτέρως σε διάφορες υπουργικές συναντήσεις και Είχα την τύχη να εκπροσωπώ και στην COP21 τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα περιβάλλοντος και πάντα είχα την αίσθηση ότι ήμουν αποδεκτός ως τμήμα της ίδιας οικογένειας. Αλλά να πω και να αναφέρω και ένα ανέκδοτο, ένα ε, περιστατικό, συγγνώμη. Όλοι ξέρουν ότι ο καθηγητής Δεμάρκο είναι ένα από τα πιο ε, δικαιωμένα πολιτικά πρόσωπα της Μάλτας, πρώην πρόεδρος της Μάλτας. Όταν συνδεθήκαμε λοιπόν κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με τον πρώην ε, ε πρόεδρο Μάριο Σουαρές σε ένα επίσημο δείπνο, Ο καθηγητής Δημάρκο με είχε συστήσει ως έναν από τους μεγαλύτερους προσπιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κόμμα μου και ένας από τα άτομα που είχαμε εργαστεί σκληρά για να εξασφαλίσουμε ότι το κόμμα μου θα τηρούσε τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Και ότι το γεγονός είναι ότι οι δράσεις μας έκτοτε έχουν καταδείξει ότι πάντα ήμασταν υπέρ του ευρωπαϊκών ιδανικών. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε και το τα φυσικά. Και αυτό καθίσταται σαφέ νομίζω, από όλε τι υπουργικέ συναντήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ πιστεύω ότι τα... οι πράξεις μιλούν πιο ηχηρά από ότι τα λόγια. Αλλά κατανοώ το ερώτημά σα και καταλαβαίνω στο πλαίσιο, το πλαίσιο στο οποίο το θέσατε και χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που είχα την ευκαιρία να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Σα ευχαριστούμε να είναι πολύ σημαντικέ οι πράξει. Γι' αυτό έθεσα το ερώτημα αυτό, οπότε σας... Έχουμε τώρα την τελευταία παρέμβαση και ο κύριος Σόλτες θα καταλήξει, θα, κάνει τις καταληκτικές παρατηρήσει. Κύριε Μπριγκάτ, λέει ο κύριος Σόλτες, σίγουρα έχετε μια μακρά πορεία και ιδίω στον ιδιωτικό τομέα και έχετε <clears throat> ιδιαίτερα να αντιμετωπίσετε οικονομικούς πόρους από διάφορες ε, πηγές. Αλλά το ερώτημα το οποίο τέθη στην αρχή αφορούσε το θέμα των εγγράφων του Παναμά και συγκεκριμένα του ρόλου που είχατε διαδραματίσει σε αυτή τη διαδικασία διακόπτει ο μιλητής. Ναι, θα μιλήσω αγγλικά, λέει ο κ. Σόλτης, αλλάζει γνώμη. Είπα ότι είναι πλούσιο το βιογραφικό σας με την εργασία σας στον ιδιωτικό τομέα και με την διαχείριση οικονομικών πόρων και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Και νομίζω ότι λαμβάνετε πολύ στα σοβαρά υπόψη και τη δική μας ε, επιμονή για τα θέματα της ανεξαρτησίας των μελών του ελεκτικού συνεδρίου. Μετά όμως και από το ερώτημα του κυρίου Σαβάρμα και βάσει άλλων πληροφοριών που έχουμε συλλέξει από, τα έντυπα, από τον έντυπο τύπο της Μάλτας σε σχέση με χιλιάδες ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία που έτυχαν διαχείρισης από το δικό σας Υπουργείο και τα οποία κονδύλια φαίνεται ότι δόθηκαν σε κάποιους συγγενείς ή κάποια μέλη του κόμματός σας και εσείς παίζετε σημαντικό ρόλο σε αυτό το πολιτικό κόμμα μετά από όλα αυτά πώς μπορείτε να εγγυηθείτε την ε, πολιτική σας ε, ουδετερότητα και αμεροληψία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη σταθερότητα και το κύρος αυτού του οργάνου. Μπορείτε να μας πείσετε ότι θα κρατήσετε αυτή την γραμμή ανεξαρτησίας για το θέμα της ανεξαρτησίας. Έχω πράγματι εμπλακεί ενεργά στον ιδιωτικό τομέα. Έχω συναντήσει και ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς λειτουργεί το σύστημα στη Μάλτα. Λένε κάποιοι πώς μπορείτε να εργάζεστε <clears throat> ως μέλος του Κοινοβουλίου στον ιδιωτικό τομέα. Στη Μάλτα, αντίθετα με άλλες ε, χώρες, τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν έχουν καν αποδοχές. Έχουν απλώς κάποια αποζημίωση. Δεν είναι πλήρους απασχόληση. Έχουμε τι οικογένειε μα που πρέπει να, να ζήσουμε. Γι' αυτό όλοι έχουν και κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν είμαστε λοιπόν ε, πλήρους απασχόλησης μέλη του Κοινοβουλίου. Όλοι είμαστε μερικής απασχόληση. Εκτός αν γίνει κάποιος από τη στιγμή που γίνεται υπουργό, τότε η μόνη πηγή εισοδήματό σου πρέπει να είναι από το λειτουργήμα αυτό. Εγώ δεν είμαι καμία εξαίρεση. Εγώ ακολούθησα ακριβώ του κανόνε που ισχύουν στη χώρα μου. Αλλά στη Μάλτα δεν είχαμε το σύστημα του πόθεν έσχες. Εγώ ήμουν ένας από τους πρώτους στο Κοινοβούλιο της Μάλτας που υπέβαλα πλήρες πόθενέσεις και πολλοί με έχουν επικρίνει γιατί συμπεριέλαβα περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω και μάλιστα για το γεγονός ότι έδινα αυτές τις πληροφορίες αμέσως, χωρίς καθυστέρηση. Όλα αυτά λοιπόν είναι πια στο δημόσιο χώρο, ακόμα και αυτά τα οποία δεν είναι μπορώ πράγματι να τα δώσω πλήρως. Ο κύριο Σόλτες αναφέρθηκε στο άλλο αυτό θέμα. Εγώ σας είπα πώς διαχειρίστηκα την Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών στη Μάλτα. Και ανέφερα και τους άλλους φορείς με τους οποίους εγώ συνεργάστηκα και έκανα σαφές ότι αυτοί οι φορείς δεν μπορούν να έχουν αξιοπιστία εάν δεν πείσουμε την κοινή γνώμη ότι πράγματι με ανεξάρτητο τρόπο λειτουργούν και με αποτελεσματικότητα. Και όταν μέλος αυτής της Επιτροπής, εργάστηκα πάρα πολύ και ακόμα και σε άλλες επιτροπές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου υπήρξα από το κόμμα μου <clears throat> σκιώδης ε, Υπουργό Εξωτερικών, πάντα τόνισα ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία στάση από όλους μας και μια συνεργατική προσέγγιση. Καταλαβαίνω ότι ο κύριο ε, Σόλτε αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Θέματα που εμπλέκουν ε, συγγενείς κτλ. Εάν καταλαβαίνω καλά αναφέρεστε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο EFRD, το Ταμείο Αγροτικών Εγγύησεων. Είναι τμήμα λοιπόν της συνολικής ευθύνης του Υπουργείου μας, η οποία όμως αντιμετωπίζεται με μια ετήσια κοινοβουλευτική διαδικασία. Εγώ δεν έχω πάρει κανένα παράπονο, καμία διαμαρτυρία για τα θέματα αυτά αυτήν μέχρι αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που ήρθαν αυτές οι καταγγελίες στη γνώση μου, όπως έκανα και σε οποιαδήποτε περίπτωση στο παρελθόν, τα παρέπεμψα στον αρμόδιο αξιωματούχο για την εποπτεία για <clears throat> πληροφορία σε σχέση με τις συγκεκριμένες δράσεις που έχουν κάνει από τη δική τους πλευρά. Και στο ενδιάμεσο διάστημα εγώ δεν είμαι στην κυβέρνηση πια και δεν ξέρω τι έχει γίνει στους τελευταίους μήνες. Υπήρξαν κάποια άθρα στον τοπικό τύπο της Μάλτας και τώρα το θέμα αυτό είναι στα χέρια της, της αυτόνομης ε, επιτροπής στην οποία δημιούργησε και στην οποία έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός τον οποίο χρησιμοποιώ πάντα όταν υποβάλλονται παράπονα και γι' αυτό το τρόπο, είμαι, είναι γαλήνια η συνείδησή μου, πάντα όταν είχα κάποιο παράνομο, παράπονο ακόμα και όταν ήταν ανώνυμες καταγγελίες για θέματα δυνητικών καταχρήσεων για την νυχθειοκαλλιέργεια, εγώ πάντα πηγαίνα στην αρμόδια ε, αστυνομική αρχή για περαιτέρω έρευνα. Δεν έχω λοιπόν κανένα πρόβλημα, ακόμα και αν αυτό αφορά κάποιο μέλος του Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβετε ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τηρηθεί η διαφάνεια. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, τέλειωσε ο χρόνος μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ε, Χαρήκαμε πολύ που σας είχαμε. Και συνεχίζουμε με την επόμενη ακροασή μας με τον επόμενο υποψήφιο. Ευχαριστώ. Uh, λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε με την τρίτη μας ακρόαση. Καλώς ορίζω τον κύριο Ζουαό Φικιουρέδο. Συγγνώμη, μας περιμένετε, καθυστερήσαμε, αλλά ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα, πολλές ερωτήσεις. Το ευαίνετε και εσείς θα δεχτείτε πολλές ερωτήσεις. Οπότε, παρακαλώ, ξεκινήστε με την εισήγησή σας. Θα ακολουθήσει ο εισηγητής, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Στην συντομή αυτή εναρκτήρια παρουσίασή μου θα μιλήσω γαλλικά και αγγλικά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εμφανίζομαι ενώπιόν σας, όμως είναι και μεγάλη ευθύνη Πρώτον, λόγω της σημασίας του Ελληνικού Συνεδρίου στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον ε, έχω επίγνωση της πολυπλοκότητας του ρόλου του Ελληνικού Συνεδρίου. Είναι επίσης ε, τεράστια ευθύνη διότι διαδέχομαι τον Πορτογάλο ε, μέλος και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Βίκτορ Καλντέιρα, ο οποίος έφερε σε πέρα με εξαιρετικό τρόπο τα καθήκοντά του και ω πρόεδρο και ο οποίο αποτελεί τιμή για τη χώρα μου. Για όλου αυτού του λόγου. θεωρώ ότι ω υποψήφιο φέρω τεράστια ευθύνη. Να υπογραμμίσω του λόγου του οποίου πιστεύω ότι αξίζω την εμπιστοσύνη σα. Θεωρώ καταρχάς ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να αποκαταστήσουμε μια σχέση η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Και Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία τη επαγγελματική μου σταδιοδρομία και να εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι μπορώ να φέρω σε πέρα στα καθήκοντά μου. Πρώτα απ' όλα εργάζομαι στη δημόσια σφαίρα εδώ και 38 έτη. Στη δημόσια διοίκηση έκανα την καριέρα μου προ το κοινό συμφέρον, γιατί αυτό ακριβώ ε, ήταν και αυτό το οποίο είχε μεγαλύτερη σημασία για μένα. Σήμερα είμαι δικαστή μέλος του Πορτογαλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ασκώ τα καθήκοντά μου εδώ και 8 χρόνια. Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφαρμόζω την ε, ισχύουσα εθνική νομοθεσία αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ήμουν ε, αρμόδιος για ελέγχου συμβατότητας συγκεκριμένα και διαπίστωνα την οικονομική ευθύνη, την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης. Επίσης έλθε την έκθεση προς τη Βουλή. Ω δικαστή, ω μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου, είχα λάβει καθήκοντα σε διάφορου τομεί και σε όλα τα επίπεδα τη δημόσια διοίκηση. Είχα ευθύνε σχεδιασμού, εκτέλεση, υλοποίηση και ελέγχου προπολογισμών, ικανού μεγέθου. Επίση, έλαβα και κυβερνητικέ θέσει στο Υπουργείο Οικονομικών ω υφυπουργό δημόσια διοίκηση δρομολόγησα σημαντικέ, θα έλεγα, πιστεύω τουλάχιστον μεταρρυθμίσει στην Πορτογαλική Δημόσια Σε αποφάσεις μερικές πολύ σημαντικέ ε, αποφάσεις για τα οικονομικά της χώρας. Μεταξύ αυτών ορισμένες αφορούν τον προπολισμό και είχα και στενές σχέσεις και συνεργασία με το Κοινοβούλιο και επιτροπές του. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να σας πω επίσης δύο λόγια σχετικά με τα κίνητρά μου. Τι με οθεί να προσπαθήσω να φέρω σε πέρα στον εαυτό ρόλο. Πιστεύω σε βάθος το ευρωπαϊκό εγχείρημα στα αρχές και τις αξίες που το διέπουν από την σύλληψή του. Με υπέρ της Ευρώπης, της ειρήνης στην Ευρώπη, την ευμερία των ευρωπαϊκών πολιτών, την ε, στιβαρή και ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών και των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει έναν ικανό πλήθος σημαντικών προκλήσεων. Είμαι πεπισμένο όμω ότι οι χώρε και οι λαοί τη Ευρώπη μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτέ τι προκλήσει αποτελεσματικά μόνο εφόσον θα είναι ενωμένοι. Κατά τη διάρκεια τη μακρόχρονη σταδιοδρομία μου, έμαθα ότι η χρηματοοικονομική διαχείριση πρέπει να είναι στο κέντρο των πολιτικών μα και θεωρώ το κράτος δικαίου πολύ σημαντικό. Όμως ταυτόχρονα θεωρώ ότι πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τον ρόλο της διαχείρισης της οικονομίας, της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων, θα είναι πιο διαφανής διαχείριση και θα υπάρχει περισσότερη λογοδοσία στα μάτια των πολιτών. Πιστεύω λοιπόν στις ε, αξίες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Συνέδριο πιστεύω στην ανεξαρτησία, την εμεροληψία, την ακαιρεότητα και την συνδελφικότητα. Αυτέ είναι οι αρχέ που διέπουν και τη δική μου δράση εδώ και πολλά χρόνια. Για μένα το έργο αυτό, στην καρδιά λοιπόν του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματο, αποτελεί τη νέα μου πρόκληση. Πιστεύω ότι χάρη στην προηγούμενη σταδιοδρομία μου είμαι έτοιμο να αναλάβω τα καθήκοντα αυτά. Είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να έχουμε περισσότερο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το βασικό μας εταίρο, και δι την Επιτροπή σας ελέγχου του προπολισμού. Πρέπει λοιπόν να εισακούσουμε τις δικές σας ανησυχίες και αιτήματα. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τον διάλογο με τα αντίστοιχα ελεγκτικά όργανα στα κράτη-μέλη. επόμενη βεβαίω την ανεξαρτησία του. Και τέλο, αυτό το οποίο αποτελεί για μένα το σημαντικότερο κίνητρο είναι να υπηρετήσω στον ύψιστο βαθμό τους Ευρωπαίους πολίτες. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για την εισηγήσή σας. Εννοείται ότι θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Ο κύριος Σαρβάμα καταρχάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Φιγκυρερό. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Στις γραπτές απαντήσεις που μας διαβιβάσατε, αναφέρετε ότι το ελεγκτικό έργο και ο προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου του ελεγκτικού συνεδρίου θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ανάλυση των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου που συνδέονται με τις ε, χρηματοοικονομικές ροές ανά τομέα ή ανά κράτος μέλος με μια κυκλική προοπτική που θα καλύπτουν και ενδεχόμενους τομείς υψηλού κινδύνου. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ φιλόδοξο, πολλά υποσχόμενο. Σας ρωτώ όμως, Πείτε μας δύο λόγια παραπάνω, καταρχάς, για την πολιτική σημασία. Για σας προσωπικά, του να υπάρχουν πραγματικά διαφανείς πληροφορίες για το πώς δαπανώνται οι πόροι των της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κρατημέλη. Και κατά δεύτερον, πόσο δεσμευμένος είστε εσείς προσωπικά για να υπάρξει Ε, απέτηση από πλευρά του Ελεκτικού Συνεδρίου για να αντιδρούνται στοιχεία βάση κράτου μέλου και βάση περιφέρεια από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κ. Πικυρίδη για να απαντήσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, Όντως, έτσι απάντησα στο ερωτηματολόγιο, στις γραπτές ερωτήσεις. Και αυτό, γιατί έχω την εντύπωση ότι αν υπάρχει μια γενική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα συστήματα ελέγχου σε όλη την Ευρώπη, έχοντας υπόψη τα συστήματα που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο σε κάθε, σε κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη το ότι υπάρχουν εξωτερικοί ανεξάρτητοι έλεγχοι εκεί και το ότι υπάρχουν και εσωτερικοί έλεγχοι, Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα και θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο θα μπορούσε να ηγηθεί της, ε, του κινήματος αυτού για την καλύτερη αξιοποίηση όλων αυτών των συστημάτων ελέγχου στην Ευρώπη. προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και να προωθηθεί και αν θέλετε μια γενική κουλτούρα οικονομίας στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να πτύξει μια προσέγγιση με τα εθνικά θεσμικά όργανα με τα ανώτατα θεσμικά όργανα ασφαλώς, αλλά και ότι βασικά τα κύρια σημεία των ιστορικών συστημάτων θα πρέπει να αξιοποιήσουν το έργο που γίνεται στο ιστορικό τους και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο αξιοποίησης των μηχανισμών αυτών στην Ευρώπη. Αν αυτό γίνει προσεκτικά με την ανάπτυξη των ίδιων μέθοδων σε όλες τις χώρες, βάσει των ίδιων αρχών, ενδεχομένως στο μέλλον να καταλήξουμε σε πιο αξιόπιστες πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού επίπεδου. Και νομίζω ότι με την απάντηση αυτή απαντώ και στο πρώτο ερώτημα που μου θέσατε για την πολιτική σημασία της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την πτυχή του κράτους μέλους. Ρωτήσατε τώρα ποια είναι η προσωπική μου δέσμευση για την ε, πρόθεση της νοοτροπίας αυτής. Εδώ ασφαλώς μπορώ να πω ότι προτίθεμαι να το κάνω αυτό. Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσω στο σημείο αυτό ότι το Ελεκτικό συνέδριο αποτελεί ένα συλλογικό σώμα. Και όσο εκ τούτου ε, υποχρεούμε να καταθέτω προτάσεις στο σώμα των ελεγκτών, να συζητώ τις προτάσεις αυτές και να περιμένω και να αναμένω τις αποφάσεις όλων των ελεγκτών. Δεν είμαι το μόνο μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Είμαι ένα μόνο μέλος. Άρα Χρειάζεται συνεργασία με τους συναδέλφους, είναι αιματικό το έργο. Και ασφαλώς και οι συνάδελφοι έχουν τη δική τους άποψη. Θα πρέπει λοιπόν να σχηματίσει το ανεξάρτητο αυτό σώμα μια ανεξάρτητη θέση. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας, αλλά αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που σας θέτω το ερώτημα αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι είναι σώμα το ρεκτικό συνέδριο, αλλά έχουμε 28 μονοκρατή μέλη και κάθε άποψη μετράει και την δική σας άποψη, την δική σας τοποθέτηση εξετάζουμε εδώ σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ρωτάω ακριβώς αυτό, τη δική σας άποψη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τον κύριο Φιγιαρέντο και να τον καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Βλέποντας το βιογραφικό του, βλέπω ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με συστήματα ε, σοφρονιστικής ε, αντιμετώπισης των ε, εγκληματιών και τέτοια θέματα. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να εφαρμόσετε αυτή την ε, πείρα που έχετε πέραν του αστείου τώρα. Σας ευχαριστώ για την εκτενή σας απάντηση και φυσικά έχετε μια σημαντική εμπειρία σε πάρα πολλούς τομείς και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, ακόμα και στο πια, στα πιο σκληρά κομμάτια, για να το πω έτσι, της πορτογαλικής ε, δημόσιας διοίκησης. Τώρα, έρχομαι στην εμπειρία σας στο Πορτογαλικό Ελεκτικό Συνέδριο. Θα ήθελα να μας πείτε με ποιο τρόπο, κατά την άποψή σας, θα μπορούσε να αναπτυχθεί η σχέση αυτή μεταξύ των Εθνικών Ελεκτικών Συνεδρίων και των κυβερνήσεών τους που είναι ελεγχόμενες οι κυβερνήσεις αυτές από τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, με ποιο τρόπο θα μπορεί βάσει τη δική σας εμπειρία δεδομένου ότι η Πορτογαλία εξακολουθεί να είναι μια χώρα του χώρα συνοχής και επομένως έχουν μεγάλη σημασία τα διαδοτικά ταμεία. Πώς νομίζετε λοιπόν θα μπορούσε να ε, εξασφαλιστεί μια πιο παιδαγωγική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών να μπορούν να υπάρχουν παραγωγικά κάποια σημεία τα οποία θα τα διευκρινίσει καλύτερα το ελεκτικό συνέδριο σε σχέση με τη λειτουργία του προπολογισμού. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια να βοηθήσουν για τη βελτίωση της εφαρμογής των ε, διαφθορτικών ταμείων από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό που σε μεγάλο βαθμό πατά για το γεγονό ότι οι κανονισμοί εκπονούνται στι Βρυξέλλε. Το μεγαλύτερο μέρο τη εφαρμογή του γίνεται στα κράτη-μέλη και από τα κράτη-μέλη. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, καλύτερη λειτουργία. Ένα. Δεύτερον, με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε την ε, χρονική υστέρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την εφαρμογή του προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών, όταν πρόκειται για προϋπολογισμούς συνδιαχείριση γιατί βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά έχουμε τις Βρυξέλλες οι οποίες εμποδίζουν την διόγκωση του δημοσίου χρέους μέσα του, μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας. Από την άλλη πλευρά, η υπογραφή των συμφωνιών για τα λειτουργικά αυτά προγράμματα δεσμεύει τα κράτη να τα χρηματοδοτήσουν. Αυτά τα δύο ερωτήματα που θα ήθελα να απαντήσετε, αν μπορείτε. Παρακαλώ. Κυρία Αγιάλα Σέντερ, σας ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Είναι πολύπλοκα τα ερωτήματά σας. Με την άδειά σας θα απαντήσω στα γαλλικά, γιατί καταλαβαίνω με τα γαλλικά, τα ισπανικά συγγνώμη, αλλά δεν τολμώ να τα ομιλήσω. Λοιπόν, με έχετε ρωτήσει πώς θα βελτιώσουμε τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν να υπομισθούν τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια για να υπάρξει μια καλύτερη χρήση των κονδυλίων αυτών. Θα σας έλεγα καταρχήν ότι λαμβάνοντα υπόψη αυτό που έχει γίνει στη χώρα μου, αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο ετέθη στην Πορτογαλία, γιατί η Πορτογαλία έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είχε πάντα αυτό το υψηλό επίπεδο απορρόφησης, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και προβλήματα σε άλλα κράτη-μέλη, εκεί που τίθεται αυτό το θέμα, με σημαντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τη συνολική χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι όταν έχουν όταν υπάρχουν κονδύλια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, αυτό εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να δώσει μια απάντηση στα νέα προβλήματα τα οποία αναδύονται. Αυτό οδηγεί σε μια κάποια ακαμψία στους ε, μηχανισμούς του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ποιος λοιπόν πρέπει να είναι ο ρόλος που θα, αναπτύξει, θα αναπτύξουν τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια για να θεραπεύσουν αυτή την κατάσταση. Αν υπενθυμίσω το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Σεβαρμά σε ένα άλλο επίπεδο. Υπάρχει ένας ρόλος, ένας χώρος έφορος για ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ελεκτρικών Συνεδρίων των Εθνικών λοιπόν ε, ελεκτρικών Συνεδρίων και του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τον πιο συγκεκριμένο τομέα της σχεδίασης των ελεκτικών δραστηριοτήτων, των δραστηριοτήτων ελεκτικού λογιστικού ελέγχου. Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κοινή σχεδίαση για να μην υπάρξει επικάλυψη και διπλή χρήση πόρων για την λειτουργία αυτή, αλλά και για να μπορέσει το ελεκτικό συνέδριο να απελευθερώσει περισσότερους υλικούς και ανθρώπινους πόρους για να μπορέσει να ε, φέρει σε πέρας άλλα εγχειρήματα και να εξυπηρετήσει άλλους στόχους. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η συνεργασία σε ό,τι αφορά την σχεδίαση των δραστηριοτήτων λογιστικού ελέγχου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και των Εθνικών Φορέων. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε, να ανοίξουμε ένα νέο χώρο για την καλύτερη χρήση των κοινωτικών κονδυλίων και κυρίως σε ό,τι αφορά το δίκτυο των ε, ανωτάτων φορέων ελέγχου πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μία ε, ιεραρχική προσέγγιση αλλά μία περισσότερο δικτυακή εν, ε, συνεργασία. Μπορεί λοιπόν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνεδρίο να βοηθήσει ορισμένους από αυτού τους ανώτατους εθνικούς φορείς να δημιουργήσουν τις κατάλληλε δομές για την καλύτερη χρήση των ε, κονδυλίων τη ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίε από τη μία χώρα στην άλλη. Δεν ξέρω τώρα αν, είχα, έχω απαντήσει στο ερώτημα που θέσατε. Για το δεύτερο ερώτημα που θέσατε για την χρησιμοποίηση των κονδυλίων σε περιπτώσει στην περίπτωση που τα κονδύλια αυτά είναι αντικείμενο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των Εθνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένας χώρος όπου μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και των Εθνικών Ελεκτικών Φορέων. Το λέω αυτό χωρίς να εννοώ ότι δεν έχει υπάρξει και στο παρελθόν προσπάθεια και πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή. Απλώς λέω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, γιατί έχω αρκετή εμπειρία στα θέματα αυτά για να ξέρω ότι <clears throat> όταν φτάνει κανείς σε ένα θεσμικό όργανο <clears throat> υπάρχει ένα παρελθόν, υπάρχουν προηγούμενες εργασίες, υπάρχει μια προηγούμενη διάγνωση ήδη για τις δυσκολίες που υπάρχουν και φυσικά γνωρίζω ότι υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ο Ντέρεκ Βον είναι ο επόμενος ομιλητής. Και πρόεδρε, ε, καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον υποψήφιο για την ομιλία του. Σας ε, Σας χαιρεπίσεις. Ε, βλέπω και ένα μεγάλο όνομα εδώ, το μεγαλύτερο από τα των άλλων υποψηφίων. Και συγχαρητήρια για το βιογραφικό σας. Νομίζω διαβάζοντας το κανείς δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία για την ανεξαρτησία και την πείρα σα σε θέματα διαχείριση και ελέγχου. Πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό. Ακριβώ επειδή είναι πολύ εντυπωσιακό το βιογραφικό σα, θα περιστώ σε μια ερώτηση που αφορά τον ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου και το ρόλο του στο μέλλον. Η Επιτροπή μας, ξέρετε, έχει συζητήσει διαμακρόν το κατά πόσο μπορούμε να μετρήσουμε, για παράδειγμα, τη συμμόρφωση. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε, να ποσοτικοποιήσουμε την απόδοση. Αυτά είναι πράγματα που μας απασχολούν και ε, από αυτό θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια. Επειδή μας είστε ακόμη περισσότερο πεπειρεμένος ελεγκτής, αν εκλεγείτε. Θα είστε ένας παραδοσιακός ελεγκτής, ο οποίος ε, θα ασχολείται μάλλον με την συμμόρφωση ή θα είστε από τους μεταρρυθμιστές, θα προσπαθείτε να μετρήσετε την απόδοση, θα προσπαθήσετε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας και δράσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για το όνομά μου Δυστυχώς ναι, στην Πορτογαλία τα ονόματα μακροσκελή έτσι ναι, στην Πορτογαλία αλλά μόνο τρία ονόματα μπορούμε να έχουμε στην ταυτότητά μα. Τέλο πάντων, στην οικογένειά μου όλοι έχουν ε, μεγάλα ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούμε το πρώτο και το τελευταίο για ευκολία όλων. Ζωάν Φιγκερέιδο, νομίζω, είναι κάτι παραπάνω πάνω από αρκετό. Αυτό χρησιμοποιώ και στη σταδιοδρομία μου. Λοιπόν, με ρωτήσετε. Τι πιστεύω πως βλέπω το μέλλον του ελεγκτικού συνεδρίου και τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Είναι μεγάλη η συζήτηση. Άλλωστε τα έχετε συζητήσει κι εσείς εδώ διαμακρών στο παρελθόν. Έχουν γίνει τόσες συζητήσεις. Διάβασα και μάλιστα θυμήθηκα και να εγγραφώ σα του 14, δεν κάνω λάθο, σχετικά με τον ρόλο στο μέλλον του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οπότε δεν ξέρω, μάλλον δεν θα πρωτοτυπήσω προκειμένου, γιατί τα έχουμε πει αυτά τα, και τα έχετε πει. Και όχι μία μόνο φορά. Δεν έχω λοιπόν πολλές καινοτόμους ιδέες, όμως επειδή με ρωτήσετε, ε, μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στην Πορτογαλική Βουλή, όταν έμαθαν ότι θα έρθω εδώ, με ρώτησαν ακριβώ για τον μελλοντικό ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Και θα σας πω τι τους είπα, τι απήντησα. Τους είπα ότι κατά πρώτον δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το ελεγκτικό συνεδρίο είναι ένα μόνο από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν συζητούμε το παρόν και το μέλλον αυτών των θεσμικών οργάνων, να μην ξεχνούμε ότι το ελληνικό συνέδριο είναι ένα εκ των πολλών. Πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα θεσμικά όργανα αυτή τη στιγμή είναι, και το λέω ως Ευρωπαίος πολίτης, γιατί αυτό είμαι αυτή τη στιγμή, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη στα μάτια των πολιτών. Αυτό αφορά και το ελεγκτικό συνέδριο. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε ότι κάτι κάνουμε και αυτό το οποίο κάνουμε έχει αξία. Αν το ελεγκτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταφέρει αυτό, να εξασφαλίσει η εμπιστοσύνη, θα έχει αποτύχει. Χρειάζεται λοιπόν να συλλέγει και να αξιολογεί στοιχεία έγκυρα τα οποία θα εμπνέουν εμπιστοσύνη στους άλλους. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνει και αυτό νομίζω ότι θέλει να κάνει το ελληνικό συνέδριο. Προς το σκοπό αυτό λοιπόν, τι μπορεί να κάνει το ελληνικό συνέδριο. Ε, είναι να βελτιώσει και την εμπιστοσύνη στα άλλα θεσμικά όργανα. Είναι μια προτεραιότητα για σήμερα, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε και τις προτεραιότητες για το μέλλον. Πρέπει να αναλογιστούμε, να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο λειτουργία μας για σήμερα και για αύριο. Και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αναθεωρούμε τους στόχους τους στρατηγικούς στόχους του 2020. Να αναθεωρούμε, να επανεξετάσουμε διαρκώς ε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ούτω καθεξής. Να επανεξετάζουμε πολιτικές για την μετανάστευση, για την ασφάλεια, την, για την οικονομική κρίση, τις μελλοντικές προκλήσεις κλπ. Για όλα αυτά λοιπόν έχω τις ιδέες μου ε, και αν θέλετε πιο συγκεκριμένα ναι, μπορώ να αναφερθώ σε έναν προϋπολογισμό εστιασμένο στα αποτελέσματα, προσανατολισμένο σε αποτελέσματα, σε απτά αποτελέσματα. Το έχει συζητήσει αυτό η Κομισιόν και νομίζω το επιδιώκει. Επίσης, το ελληνικό συνέδριο πρέπει να υποστηρίξει κάθε κίνηση, κάθε δράση τη Κομισιόν προς ένα καλύτερο και πιο ευέλικτο πλαίσιο δημοσιονομική διαχείριση, με πιο ευέλικτου κανόνε. Ένα πλαίσιο που θα αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες, τις πραγματικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συγκεκριμένες δράσεις της Κομισιόν. Μετά υπάρχουν και άλλες ε, δράσεις που έχουν σχέση με το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο. Για παράδειγμα, έχουμε το ζήτημα της αξιολόγησης και βελτίωσης της αποδοσής μας. Έχουμε τα ας το πούμε, νέα προϊόντα. Για παράδειγμα, εκτός από τις ε, ειδικέ, έχουμε και τις γενικές εκθέσεις. Πρέπει να έχουμε και γενικές εκθέσεις. Ε, πρέπει να βελτιώσουμε την ταχύτητά μας. Είναι θέμα το οποίο έχετε συζητήσει και εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Να ενισχύσουμε τον διάλογο με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να συζητήσουμε το θέμα του σχεδιασμού των ελέγχων κλπ. κλπ. Αυτά όμως τα γνωρίζετε. Είναι ιδέες που είναι στο μυαλό το δικό σας αλλά και των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Εάν ε, εγκρίνετε την υποψηφιότητά μου και εφόσον ε, διοριστώ, αυτή είναι και η στόχη του οποίου θα επιδιώξω. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ιδέες σας. Είναι εντυπωσιακή η επαγγελματική σας εμπειρία γιατί έχετε βρεθεί και ένθεν και ακήθεν των οδοφραγμάτων το είπιν και επομένως είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς μπορεί να συνδυάσει αυτές τις δύο πτυχές εμπειρία σας για τα θέματα ελέγχου. Επειδή όμως πρέπει να περάσουμε στη πληροφορία, θα ζητήσω από τον κύριο Σόλτες να κλείσει και ίσως αν θέλει να θέσει και άλλα ερωτήματα Ευχαριστώ. Ήταν πολύ εντυπωσιακή η παρουσίασή σας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ε, ικανότητά σας και για την κατανόηση που έχετε δείξει της προβληματικής και των ε, προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσετε να μεταλαμβαδεύσετε και κάποιες βέλτιστες πρακτικές από το Τριμπουνά του Σκόντους στην Πορτογαλία και στο Ευρωπαϊκό ε, Ελεκτικό Συνέδριο. Βέβαια δεν είναι το ίδιο σαν να είναι κανείς δικαστικός εκεί, αλλά σίγουρα νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να ενισχύσουμε ενδεχομένως και τις εξουσίες αυτού του φορέα ώστε να έχει και κάποιο κομμάτι από το χαρακτήρα ενός πραγματικού δικαστηρίου γιατί η λογοδοσία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και τέλος, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε καλύτερα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και να ενισχύσουμε το κύρος του ώστε οι συστάσεις του και οι αιτήσει που περιλαμβάνονται στι εκθέσει ελέγχου να λαμβάνονται επιτέλους. Υπόψη με ένα σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, για τι απαντήσει που μα δώσατε. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, ναι, παρακαλώ. Ναι. Είπα στην αρχική μου παρέμβαση ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ ενώπιόν σα, Φυσικά εσείς είσαστε αρμόδιοι να πάρετε την απόφαση, είσαστε βουλευτέ εκλεγμένοι από τους λαούς τη Ευρώπης, θα ψηφίσετε για το θέμα της εντολής μου. Εγώ φυσικά θα αποδεχτώ την τιμιγορία σα. και θέλω να πω ότι είναι τιμή για μένα να είμαι εδώ και να έχω τύχη ερωτήσεων από ένα βουλευτή, ο οποίος και αυτός υπήρξε πρόεδρος ενός εθνικού φορέα ελέγχου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω σε όλους οι οποίοι δεν ψηφίζουν, δεν είναι βουλευτές, δεν είναι συνεργάτες, δεν είναι... Ε, αρμόδιοι για να είναι παρόντε. Ζήτω να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών ώστε να μπορέσουμε να, να περάσουμε στην ψηφοφορία για να αποχωρήσουν αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να είναι παρόντε και μετά θα κάνουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ να είστε σίγουροι ότι έχετε τι ηλεκτρονικέ σα κάρτε γιατί θα προχωρήσουμε στην ηλεκτρονική.